Bene, Αρχίζει η συνεδρίαση. Να καλωσορίσω προσωπικά την Υπουργό Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπέθρου, την κυρία Μέτε Κέρσκοφ, η οποία είναι Προεδρεύουσα του Συμβουλίου Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι Μέτε που ήρθες για να μας παρουσιάσεις το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας, ένα πρόγραμμα που έρχεται σε μια σταυρική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Ξέρουμε ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της Δανέζικης Προεδρίας το θέμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και ξέρω ότι θα συνεργαστούμε στενά για το θέμα. Έχουμε και άλλα ζητήματα Έχω κατά νου το θέμα της ευθυγράμμισης, έχουν προχωρήσει πολύ και αυτό λόγω της εξαιρετικής δουλειάς της Πολυελλονικής Προεδρίας που ελπίζουμε να συνεχίσουμε, όπως επίσης και το πακέτο για την ποιότητα και τα άλλα ντοσιέ. Σε ευχαριστούμε Υπουργέ που είσαι εδώ. Σου δίνω το λόγο λοιπόν ευθύ αμέσω για την τοποθέτησή σου. Ευχαριστώ. Μέτε. Δεύτερη, δεύτερη μέρα μου, χθε και σήμερα στο ε, Συμβουλίο το πρωί, τώρα εδώ, βέβαια είναι η συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και μιας και είμαι και νέα στη δουλειά αυτή, θα, έπρεπε θα πρέπει νομίζω να σας συγχαρώ και εσάς γιατί επανεκλεγήκατε. Δεν είσαστε βέβαια νέος, έχετε πολλή γνώση του, των θεμάτων και εγώ βεβαίως έχω μέγα σεβασμού για όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται εδώ ε, και που είναι φορείς γνώσεων και πληροφοριών για τα όσα προτίθεμεθα να αποφασίσουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε. Είμαι υπουργό Γεωργίας και άρα αρμοδία για να κάνω να προχωρήσουν τα πράγματα τη μεταρρύθμισης τη κοινή αγροτική πολιτική. Να γίνει δηλαδή η γεωργική πολιτική πραγματική. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου. Πρέπει να το κάνω στο Συμβούλιο σε συνεργασία με άλλου 26 συναδέλφου και βεβαίως και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που μπορώ να διεξαγάγω διάλογο και σε όλη τη διάρκεια αυτή με εσά εδώ στο Κοινοβούλιο, διότι αυτό που κάνουμε είναι να φτιάχνουμε την ιστορία, δημιουργούμε ιστορία. Θα χρειαστεί να με βοηθήσετε, διότι θα πρέπει να λάβουμε από κοινού αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, για πρώτη φορά τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση στην ΚΑΠ, που θα χρειαστεί να συνεργαστούμε για να βρούμε κοινέ λύσεις και ένα κοινό έδαφος. Χαίρομαι που στη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για το οικοδόμημα που θα αποτελέσει την μελλοντική και αγροτική πολιτική της Ένωσης. Θα φτιάξουμε λοιπόν τα θεμέλια αυτά ως αληθινοί γείτονε σε συνεργασία Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και αναμένω με ιδιαίτερη ανυπομονησία και ενδιαφέρον τη συνεργασία αυτή. Πρώτα θα σας ε, υποβάλω ορισμένα σχόλια, ορισμένε παρατηρήσει για τη Δανική Προεδρία και για τους στόχους μας. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια δυναμική, πράσινη και ασφαλή Ευρώπη, να είναι προετοιμασμένη και οικονομικά και κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Η Δανική Προεδρία θα καταθέσει μια ημερήσια διάταξη προενεργή για την βιώσιμη ανάπτυξη ανάπτυξη χωρίς υπερβολική χρήση των υφιστάμενων φυσικών πόρων. Είναι δύσκολο, αλλά είναι κατορθωτό. Θα προωθήσουμε την πράσινη ανάπτυξη, που αυτό είναι απαραίτητο να το δούμε ως πρόκληση και είναι απαραίτητο για τη μελλοντική ευημερία, για την ανάπτυξη και για την απασχόληση στην Ευρώπη. Βέβαια, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε αποδοτικές λύσεις και να λάβουμε υπόψη και την ανάγκη αύξηση ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ο Ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση τη πράσινη ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπω άλλωστε η κοινή αγροτική πολιτική έπαιξε σημαντικό ρόλο για το χτίσιμο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε την αγροτική πολιτική πραγματικά στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε μια πολιτική στραμμένη και κατάλληλη για το μέλλον. Από τον περσινό Οκτώβριο η συζήτηση επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση έχει παίξει κέριο ρόλο και στη συζήτηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της αναδιαμόρφωσης της κοινή αγροτικής πολιτικής και προσαρμογής της στις, στις ε, ανάγκες, προτεραιότητες και προσδοκίες των Ευρωπαίων αγροτών, πολιτών και φορολογουμένων που αλλάζουν συνεχώς. Στο χθεσινό Συμβούλιο συζητήσαμε την οργάνωση της κοινή αγοράς. Τους επόμενους μήνες θα διεξαχθούν και άλλες συζητήσεις στο επίπεδο του Συμβουλίου Υπουργών για όλες τις προτάσεις της δέσμης των μεταρρυθμίσεων. Και θα συνεχιστεί βέβαια και η τεχνική εργασία. Είναι λοιπόν πρόημα ακόμη να μπω σε λεπτομέρειε, κύριε Πρόεδρε, για τα θεμελιώδη στοιχεία τη μεταρρύθμιση. Για όλα πάντω τα πολιτικά θέματα, το Συμβούλιο όπω και το Κοινοβούλιο έχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνει. Και γνωρίζουμε ότι οι θέσει μα για ορισμένα θέματα εξαρτώνται από τι τελικέ παραμέτρου που θα ε, λάβει ο μιλωτικό προπολογισμό τη Ένωση. Ωστόσο ελπίζω ότι θα μπορέσει να ολοκληρώσει το Συμβούλιο τις πρώτες του εργασίες τον Ιούνιο με την υποβολή εκθέσεως πρόοδου. Τώρα, έχω τέσσερα γενικά σημεία που θέλω να συζητήσω σήμερα μαζί σας. Πρώτο, είναι σημαντικό να απλοποιηθεί η κοινή αγροτική πολιτική, να απλουστευτεί. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερη περιπλοκότητα, ούτε περισσότερη γραφειοκρατία. Δεύτερο, θα ήθελα να αποδώσω ιδιαίτερη έμφαση στο στοιχείο του greening, του πρασινίσματος, αν με επιτρέπετε να το πω έτσι στα ελληνικά. Είμαι βεβαία ότι το στοιχείο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο συζητήσεων. Πιστεύω όμως ακόμη ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτό το πρασίνισμα είναι στην ουσία το μέλλον. Εκεί θα αναπτυχθούν οι δουλειές, εκεί θα αναπτυχθεί η εξαγωγή. Χρειάζεται επίσης να έχουμε θετική συμβολή για να σφυριλατήσουμε μεθόδους παραγωγής οι οποίες θα επιτρέψουν προστασία του περιβάλλοντος και καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Χρειαζόμαστε καινοτομία, να δημιουργήσουμε νέες πηγές προσόδων και να έχουμε επιτυχία στις ε, αγορές εξαγωγών. Τέταρτο, θα ήθελα να αναφερθώ στην ε, διακόπτη. Θα μου δώσετε μία στο κεφάλι με το σφυρί αυτό, αγαπητέ φίλε. Τρόμαξα για μια στιγμή. Ίσως έκανα κάτι κακό, κάτι που δεν επιτρέπεται. Είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι εδώ σε Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δεν έχω συνηθίσει αυτό με τα σφυριά. Θα είμαι προσεκτική λοιπόν εδώ. Ούτε πρόκειται να χρησιμοποιώ υβρεολογίες, μη φοβάστε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε μια συνοχή πολιτικών και την άνοιξη θα διεξαχθεί η διάσκεψη των ΗΠΑ Ρίο Συν που θα εγκύψει σε ορισμένα από τα θέματα αυτά και σε άλλους τομείς πολιτικής της Ένωσης, κυρίως του εμπορίου και της ανάπτυξης. Άρα χρειαζόμαστε συνοχή των πολιτικών αυτών. Η δέσμη των μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνει και δύο μικρότερες προτάσεις. Το παραδοσιακό ε, πρόγραμμα απευθείας πληρωμών και το ε, πακέτο προσαρμογής του κρασιού για να μπορέσουν να υιοθετηθούν έγκαιρα τα νομοθετήματα αυτά, θα πρέπει ε, να τις εγκρίνουν οι συνομοθέτες το δυνατόν συντομότερο. Το Συμβούλιο είναι έτοιμο να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Και είμαι βεβαία ότι και εσείς θα συμφωνείτε με το στόχο αυτό. Τώρα για την ευθυγράμμιση της αγροτικής νομοθεσίας με την συνθήκη της Λισαβόνας. Όλα τα θεσμικά όργανα, το γνωρίζω, έκαναν μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλίσουν δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για τα οριζόντια θέματα. Ελπίζω ότι όλοι θα μπορέσουμε τώρα να κάνουμε την τελευταία απαραίτητη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια πραγματική οριζόντια προσέγγιση που θα μας επιτρέψει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στι προτάσεις μεταρρύθμισης της αγροτικής πολιτικής για θέματα ευθυγράμμισης των απότατων περιοχών μικρών νησιών του Αιγαίου και της βιολογικής παραγωγής. Θέλουμε να κάνουμε ταχεία πρόοδο έτσι ώστε ο πρώτος τριμερής διάλογος να γίνει ήδη τον επόμενο μήνα. Εδώ η οριζόντια προσέγγιση στην ευθυγράμμιση της Λισαβόνας θα είναι μέγα πλεονέκτημα. Έρχομαι και με λίγα λόγια στα άλλα ντοσιέ που συζητούνται ήδη στα θεσμικά μας όργανα, αρχίζοντας με την δέσμη μέτρων ποιότητας τροφίμων. Αυτό το δοσιέ έχει μεγάλη σημασία για τον Ευρωπαίο πολίτη, ο οποίος αποζητεί την ε, ποικιλία και την ποιότητα της αγροτικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά επιθυμεί να ενισχύσει η Προεδρία, ενισχύοντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των γεωργών της Ένωσης. Το πρώτο μισό του 2012 η Κομισιόν αναμένεται να καταθέσει έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού του 2007 για την ε, βιολογική παραγωγή που θα δώσει την ευκαιρία και στα δύο θεσμικά μας όργανα να συζητήσουμε ακριβώς αυτό το θέμα της βιολογικής παραγωγής. Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή για να καταθέσουμε τις απόψεις μας για το μέλλον της ε, βιολογικής παραγωγής στην οποία οι Ευρωπαίοι αγρότες μπορούν να βρουν ευκαιρίες για την παραγωγή προϊόντων που θα έχουν υψηλή ποιότητα αλλά και υψηλή αξία. Ακολουθεί ένα θέμα το οποίο θεωρούν πολύ σημαντικό και τα δύο θεσμικά μας όργανα, δηλαδή η ευημερία των ζώων. Μια σημαντική πτυχή του ντοσχέ αυτού θα εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της Προεδρίας. Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ο Επίτροπος Νταλή υπέβαλε έκθεση στους υπουργούς για την προστασία των ζώων στη διάρκεια της μεταφοράς των. Και όταν μιλούμε για μεταφορά ζώων, ας μην λησμονούμε ως πολιτικοί ότι οι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα εκατομμύριο πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαν στην ιστοσελίδα και υπέγραψαν για την, και ζήτησαν τη μέγιστη δυνατή προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των. Αναμένουμε επίσης να εξετάσουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και ευημερία των ζώων Γνωρίζω ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είσαστε ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς στη συζήτηση της έγκρισης της, ε, του ψηφίσματος ιδίας πρωτοβουλίας της 5ης Μαΐου 2010 για την αξιολόγηση του σχεδίου δράσεως 2006-2010 για το θέμα αυτό. Μαζί λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οργανώσουμε διάσκεψη για την ευημερία των ζώων στις 29 Φεβρουαρίου και 1 η Μαρτίου του 2012 ρίχνοντας ιδιαίτερα το βάρος για την ευημερία των ζώων, επιβολή των μέτρων και, την, και τα επιστημονικά δεδομένα. Και θα προσπαθήσουμε να συντονίσουμε την ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου μάλλον, στην ε, πρόταση της Επιτροπής για, τα, για την καταπολέμηση των μικροβίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του ότι δεν μπορούν πλέον, δεν τους πιάνουν πλέον τα αντιβιωτικά. Θα εξετάσουμε το θέμα από μια ολιστική άποψη, περιλαμβάνοντας και τον κτηνιατρικό τομέα και τον τομέα της ανθρώπινης υγείας. Έτσι λοιπόν κύριε Πρόεδρε επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω βεβαιώνοντάς σας ότι η Ιδανική Προεδρία θα πράξει ό,τι μπορεί τους επομένους μήνες ώστε να επιτρέψει τη διεξαγωγή υγιού διαλόγου μεταξύ των δύο θεσμικών μα οργάνων. Θα είμαι διαθέσιμη για τον διάλογο. Όλο μου το προσωπικό του το είπα. Το είπα στο Υπουργείο μου σε όλου και όλες. Τους είπα φιλήστε το boyfriend, φιλήστε την σύζυγο το, τα Χριστούγεννα και θα του ξαναδείτε το καλοκαίρι. Σα το λέω για να σα εξηγήσω ότι είμαστε εδώ, είμαστε πανέτοιμοι και πανέτοιμε και για τον διάλογο και ο τίτλος της δανικής μας προεδρίας είναι «Η Ευρώπη ανασκουμπώνεται» και ελπίζω ότι όντως θα δεχτείτε να το κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Υπουργέ, η παρουσίασή σου μας δίνει τη δυνατότητα για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ και τον Υπουργό Αλετράρη, τον Υπουργό Γεωργίας της Κύπρου, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικός αυτός ο δεσμός μεταξύ των δύο προεδριών, της Δανέζικης και της Κυπριακής που θα ακολουθήσει. Ξεκινάμε με τους συντονιστές. Ο Άλμπερντες έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήλθατε κυρία Υπουργέ στην Επιτροπή Γεωργίας. Είχαμε ήδη την ευκαιρία ε, να σας γνωρίσουμε και να συνομιλήσουμε μαζί σας στο μεσημεριανό γεύμα με τους συντονιστές. Η πολιτική μου ομάδα σας καλωσορίζει. Αναμένουμε με ιδιαίτερη ε, χαρά την συνεργασία στο επόμενο εξάμεινο. Θέσατε ορισμένα θέματα, θα είμαι και εγώ πολύ σύντομος και θα ήθελα έτσι να μπορέσω να δώσω τη δυνατότητα και στους συναδέλφους μου να μιλήσουν. Μιλήσατε για το πρασίνισμα. Κοιτάζω αυτό το κατάλογο. Τι έχουν κάνει για το πρασίνισμα, δηλαδή οι χώρες μέλη που κυρίως έχει χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια αυτή από τον δεύτερο πυλώνα. Εξετάζω τον πίνακα των 27 χωρών μελών και βλέπω ότι η ε, Δανία είναι η τελευταία από τους 27 διαθέτοντας λιγότερο από 40 ευρώ ανά εκτάριο στον δεύτερο πυλώνα. Ιταλία 113, Αυστρία 167 ευρώ, Σλοβενία 270 ευρώ. Δεν υπάρχουν λοιπόν μεγάλες διαφορές μόνο στον πρώτο πυλώνα αλλά και στον δεύτερο πυλώνα. Και Στη Βαβαρία είμαστε επίσης γύρω στα 200 ευρώ χρηματοδότηση ανά εκτάριο για το πρασίνισμα. Αυτό σημαίνει ότι εσείς ως πρόεδρος του Συμβουλίου θα έχετε την ευθύνη να μειωθούν οι διαφορές. Βέβαια, εσείς είστε υπουργός γεωργίας της χώρας σας εδώ και πολύ λίγο χρόνο, αλλά σημειώνω ότι η Δανία έχει κάνει τα λιγότερα από όλους. Εκεί όπου θα σας υποστηρίξω και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Άλλωστε στην έκθεσή μου, που είναι έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλέον, υπάρχει ένα ερυθρό νήμα το οποίο διασχίζει ολόκληρο το κείμενό μου και είναι η γραφειοκρατία. Διακομματικά ήμασταν σύμφωνοι ότι θέλουμε να σώσουμε τους αγρότες από τη γραφειοκρατία καθώς και τις διοικήσεις. Δεν θέλουμε να τους φορτώσουμε περισσότερη γραφειοκρατία. Είμαι πεπισμένος ότι θα σας βρούμε στο πλευρό μας στον αγώνα αυτό για τη δημιουργία δηλαδή απλοποιημένων διαδικασιών στην Ευρώπη ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χωρίς πολλή γραφειοκρατία. Γνωρίζουμε όλοι βεβαίως πόσο τεταμένη είναι δημοσιονομικά η κατάσταση. Ως Επιτροπή Γεωργίας δεν έχουμε την ύβρη να ζητήσουμε ακόμα περισσότερα χρήματα. Είπαμε ότι θέλουμε τουλάχιστον τα ίδια με τα χρήματα που είχαμε μέχρι τώρα στη διάθεσή μας. Δεν αποκλείεται βέβαια εν τέλει να μας δοθούν ακόμα λιγότερα κονδύλια. Ας το έχουμε υπόψη αυτό. Και αν, αν εν τέλει μας περικόψουν τα κονδύλια κατά 10% οι γεωργοί πλέον δεν θα, δώσουν, δεν θα έχουν απολύτω καμιά κατανόηση αν από αυτά τα περιορισμένα κονδύλια το 30% πηγαίνει στη γραφειοκρατία. Σε όλα αυτά μέσα δεν πρέπει να λησμονούμε για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας και της αποδοτικής γεωργίας. Και πιστεύω ότι ως Δανέζα υπουργό θα επιθυμείτε να παραμείνει ανταγωνιστική και η δανική γεωργία και να δώσετε το παράδειγμα και στις υπόλοιπες 26 γεωργίες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Χαίρομαι και μας είπατε άλλωστε και στη διάρκεια του γεύματος ότι θα συνεργαστείτε μαζί μας στο πνεύμα των συνθήκων, ε, στο, θα συνεχίσει μαζί μας στο πνεύμα της συνθήκης Λισαβόνας, το ίδιο καλά όπως έπραξε και ο προκάτοχός σας Πολωνός Υπουργός. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την διαθεσιμότητά σας αυτή. Ευχαριστώ Άλμπερο Λουίς Κάπουλα Σάντος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω διότι μπορέσαμε ανεπίσημα και διάρκεια του γεύματος να τα αλλάξουμε. Πώς και πρέπει να πω ότι ήταν η δεύτερη συνάντησή μας αυτή και με μεγάλη ικανοποίηση σημειώνω ότι είσαστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε εκ του σύνεγγης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίσημο επίπεδο ή άτυπα. Και θέλετε να μας συναντήσετε και πάλι όποτε επιθυμούμε. Θέλω να σας συγχαρώ διότι είναι φιλόδοξο αλλά σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλό το πρόγραμμά σας για την ε, δική σας ε, ε, προεδρία. Μακάρι να μπορούσαμε όλα αυτά να τα συγκεράσουμε ως απόψεις και να έχουμε μια ανταγωνιστική ευρωπαϊκή γεωργία με σεβασμό στο περιβάλλον έτσι όπως το περιγράφετε. Θα δω κατά πόσο θα μπορέσουμε κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας κάποιους από τους στόχους που έχετε θέσει να τα υλοποιήσετε. Και ήθελα τώρα να σας πω το εξή. Πιστεύω ότι υπάρχουν δύο ή τρία βασικά θέματα για τα οποία είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε συμφωνία πολιτική επί της αρχής μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου το συντομότερο δυνατό. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το θέμα του προπολογισμού. Θέλω να πω, για σας, για την Προεδρία. Ο προπολογισμό που προτείνει η Επιτροπή είναι ικανοποιητικός ή όχι. Δεύτερο ερώτημα. Λεπτό και πάρα πολύ πολύπλοκο. Είναι το θέμα της, επαν... της ε, αποκατάστασης της ισορροπίας μεταξύ των κρατών μελών. Και εγώ, όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, είναι απαραίτητο να κάνουμε μία προσέγγιση σφαιρική των δύο πυλώνων, διότι είναι πολύ πιο εύκολο να επαληθεύσουμε πού υπάρχουν ε, θέματα τα οποία είναι άδικα για κάποιους, αλλά αν υπάρχει τελικά ισορροπία. Υπάρχουν χώρε οι οποίε αδικούνται με κάποια θέματα στον πρώτο πυλώνα, αλλά ε, δικαιώνονται με κάποια θέματα στο δεύτερο. Θα πρέπει λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν δεν είναι πάρα πολύ φιλόδοξα, διότι λέγουν κάποια εδώ και χρόνια ότι υπάρχουν διάφορε ε, αδικίες στην ΚΑΠ σε επίπεδο κρατών, περιφερειών και προϊόντων. Τώρα λοιπόν έχουμε την μεγάλη ευκαιρία στα πλαίσια μεταρρύθμιση να διορθώσουμε αυτέ τι αδικίε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε σε σχέση με αυτά τα προτείνει η Κομισιόν τι μπορούμε να κάνουμε. Μα προτείνει ένα παράρτημα με κάποια κονδύλια για κάθε κράτος μέλο και αν δεν υπάρχει πρώτερη συμφωνία ο κάθε βουλευτής για τη χώρα του σε κάθε σημείο θα προτείνει αύξηση. Θα ανοίξουμε έτσι λοιπόν το κουτί της Πανδώρας. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μην καταλήξουμε σε νικητέ και ιτημένου, να κάνουμε κάτι που θα βοηθήσει όλου να προχωρήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε μαζί μας ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μία φόρμουλα που θα μας οδηγήσει στο να κάνουμε ε, πραγματικά κάτι δίκαιο για όλους. Πείτε μας αν είστε διατεθειμένοι να το κάνετε Τώρα το τρίτο θέμα είναι αυτό το περίσφημο πρασίνισμα. Είμαστε βεβαίως υπέρ του πρασίνισματο τη γεωργίας. Το ερώτημα είναι πώ γίνεται κάτι τέτοιο. Πείστε, πείτε μας λοιπόν σύντομα, σε γενικέ γραμμέ, τι σκέφτεται να κάνετε. Πρέπει να αλλάξουμε κάποια από τα γενικές μας αρχές ή ριζοσπαστικά να τα αλλάξουμε όλα. Ευχαριστώ. Ο George Λάιον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας Καλωσορίζω κυρία Υπουργέ. Λυπούμε που δεν ήμουν να παρόν στο γεύμα. Συνάδελφος από την Σουηδία ήταν στη θέση μου. Ξέρω ότι πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, διότι βλέπω ότι υπάρχει αίσθημα φιλίας μεταξύ και του Υπουργού και ημών. Πολύ καλύτερα λέω πήγαν τα πράγματα από ό,τι με την προηγούμενη Πολωνική Προεδρία. Άρα πρέπει να φάγατε εξαιρετικά καλά το μεσημέρι για να είναι τόσο καλέ οι σχέσει σα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να χαιρετήσω την προτεραιότητά σα για την ε, ε, αηφόρο και πράσινη ανάπτυξη της γεωργίας. Είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει πρασίνισμα, απλοποίηση και νομίζω ότι αυτά είναι αμοιβαίως ε, ε, συνδεδεμένα μεταξύ τους και συμβατά. Δεν χρειάζεται να σα πει κάτι τέτοιο. Και βεβαίω χρειαζόμαστε νέε μεθόδου, καινοτόμε μεθόδου παραγωγή των γεωργικών προϊόντων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον. Βλέπουμε ποιε είναι οι απόψει σα και στην ομάδα μου συμφωνούμε και θέλουμε να συνεχθούμε μαζί σα. Ξέρουμε ότι είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση με την Πολωνική Προεδρία, είδαμε τον Υπουργό πάρα πολλές φορές και έτσι μπορέσαμε κάποια από τα θέματα που μας απασχολούσαν στην πρόταση της Επιτροπής να διευκρινίσουμε και ελπίζω ότι και την τη της δικής σας Προεδρίας θα συνεχίσει να υπάρχει σε αυτόν τον τομέα Πρόεδρος. Κατά την άποψή σας, πώς πιστεύετε ότι θα προοδεύσουν τα πράγματα. Στο MFF πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία, δεδομένου ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μεταρρύθμιση της κάποιες αποφάσεις που ληφθούν. Εμείς είμαστε της απόψη ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για καμία μεταρρύθμιση αν δεν ξέρουμε ποια είναι η τελική άποψη για το MFF. Δηλαδή δεν ξέρουμε, αν δεν ξέρουμε πόσα κονδύλια θα έχουμε στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να κάνουμε ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Κατά την άποψή σας, δεδομένου ότι υπάρχουν και εκλογέ σε πολλέ ευρωπαϊκές χώρε που καθυστερούν τα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση κάτι τέτοιο να προοδεύσει. Επίσης, το θέμα τη ευημερία των ζώων είναι κάτι που μας απασχολεί εμά. Το ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση ε, για την Ευρώπη σε κάποιες χώρες για την συστοιχία κλοβών και ξέρουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν κότες που γεννούν αυγά όχι σε κανονικέ συνθήκε και παρόλα αυτά τα αυγά αυτά διοχετεύονται στις ευρωπαϊκές αγορές. Τι σκέφτεσαι να κάνετε με τις χώρες αυτές, με τους παραγωγούς αυτού. γιατί ξέρω ότι πάρα πολλέ φορές, ε, και λέγεται αυτό, έχουν επενδυθεί εκατομμύρια για να συμμορφωθούν όλοι οι πτηνοτρόφοι με τις ε, ευρωπαϊκές υγείες, αλλά δεν έχουν γίνει ε, τα πράγματα σωστά. Τι κάνετε λοιπόν με την εκπνοή της συμμόρφωσης που είναι για φέτος τον Ιανουάριο. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση έως το τέλος του χρόνου. Επίσης, ξέρουμε ότι σε πολλές χώρες από μας δεν έχει επιτευχθεί η συμμόρφωση και μας ενδιαφέρει να μας πείτε τι θα κάνετε. Πιστεύουμε ότι κάποιοι δεν θα μπορέσουν να σεβαστούν τις προθεσμίες που έχουν τεθεί. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι του χρόνου τον Ιανουάριο θα πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να μπορέσει να υπάρξει πρόοδο σε αυτόν τον τομέα, γιατί, όπως σας είπα, με ενδιαφέρει αυτό το θέμα τη ευημερία των ζώων γενικότερα και των πτηνών. Ευχαριστώ και πάλι, σας συγχαίρω και είμαι στη θέση σα για συνεργασία αγαστή μαζί σας. Ευχαριστώ, κύριος Νίκολσον. Με ευνηδιάσατε λίγο. Ορισμένα από τα θέματα που θέλω να πω έχουν ήδη καλυφθεί και θα καλυφθούν κι άλλο βέβαια, κυρίως ο προπολογισμό είναι το μείζον. Και μέχρι ότου έχουμε τον προϋπολογισμό, κανένα μας δεν μπορεί να μαντεύσει το μέλλον. Ένα άλλο θέμα είναι η αστάθεια των αγορών. Και τι γίνεται. Εγώ ήμουν εισηγητής για τα γαλακτοκομικά. Το ζήτημα είναι τι γίνεται, διότι μπορούμε να ελέγξουμε την παραγωγή, μπορούμε να ελέγξουμε τη μεταποίηση, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ωστόσο το λιανικό εμπόριο. Και εκεί όσο δεν μπορούμε, αυτό θα οδηγεί σε αστάθεια των αγορών. Εγώ πιστεύω όντως στην απλότητα. Σας το έχω ξαναπεί, αλλά θα το ξαναπώ. Και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν πιστεύω όμως ότι αν βάλετε στον πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα το πρασίνισμα ότι θα μπορέσετε ε, να πάτε στην απλότητα και στη μείωση γραφειοκρατίας. Άκουσα τον Τζόρτζ να λέει ότι γίνεται. Αναμένω να δω πώς. Εάν όμως το βάλετε στον πρώτο πυλώνα όπως είπα θα έχετε περισσότερο έλεγχο, περισσότερες επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αγροκτήματα και ούτω καθεξής. Δεν θα πρέπει να γίνεται επιθεώρηση στα αγροκτήματα παραπάνω από μια φορά το χρόνο και θα πρέπει να γίνεται όλο μαζί μια φορά, όλα δηλαδή, one stop shop και να ξεμπερδεύουν μετά οι γεωργοί. Είμαστε ήδη στα μέσα του Γενάρη Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και έχουμε τα σχετικά νούμερα. Να συνεχίσει ωστόσο να ασκείται πίεση σε αυτούς που οφείλουν να τα εφαρμόσουν τα μέτρα. Μη λησμονούμε ότι η νομοθεσία έχει εγκριθεί από τη σκοπιά της προστασίας των ζώων. Και όχι από την πλευρά των καταναλωτών, που αυτό που θέλουν είναι η παραγωγή να είναι ε, τέτοια που να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες προστασίας των ζώων. Και τώρα για το κεφάλαιο 14 και της μεταρρύθμισης. Εξακολουθούμε να εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ευρωπαϊκές χώρες, τεράστιες ποσότητες τροφίμων που παράγονται σε χώρες οι οποίες ουδέμια σχέση έχουν με τα πρότυπα παραγωγής τα δικά μας ή της προστασίας των ζώων ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως κλείνουμε τα μάτια και εξακολουθούμε να επιτρέπουμε τις εισαγωγές αυτές και να αναγκάζουμε τους δικούς μας παραγωγούς να αγωνίζονται, να ανταγωνίζονται κατά των άλλων με το ένα χέρι δεμένο από την πλάτη. Γι' αυτό και λένε οι αγρότες ότι η κοινή αγροτική πολιτική δεν λειτουργεί υπέρ μας. Αυτό είναι μια δυσκολία που έχουμε. Ορισμένοι Ανησυχούμε πάρα πολύ, αγαπητή κυρία Υπουργέ, όταν βλέπουμε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις από πλευράς Ένωσης με τις χώρες Μερκοσούρ. Πού μπορεί να καταλήξουν. Εγώ ήμουν από τους ανθρώπους που πήγαμε στη Βραζιλία προπενταετίας περίπου και όταν επιστρέψαμε και ζητήσαμε και είπαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι σωστά τα συμπεράσματά της. Πολύ σύντομα απαγορεύτηκαν οι εισαγωγέ βραζιλιανού βόηου κρέατο διότι δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα τα δικά μας. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει και σε πολλούς άλλους τομεί τη παραγωγής των χωρών εκείνων. Και οι γεωργοί μας δεν κατανοούν πλέον γιατί επιτρέπουμε να γίνεται αυτό. Αυτό είναι απαράδεκτο και ασφαλώς τους βλάπτει. Και δεν το καταλαβαίνουν, δεν κατανοούν οι, αγρότε αγρότες γιατί εξακολουθούμε να κλείνουμε τα μάτια. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στο έργο σας, στο επόμενο εξάμεινο που θα είναι δύσκολο. Και όπως είπατε στην αρχή, οι συνεργάτες και οι σύμβουλοί σας δεν θα έχουν και πολύ χρόνο ελεύθερο στη διάθεσή τους, γιατί θα έχουν πολλά, πράγματα, πολλά θέματα να χειριστούν. Ευχαριστώ. Χόισλινγκ. Και εγώ, κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι καλή επιτυχία για το επόμενο εξάμεινο. Ευτυχώς για σας είναι μόνο έξι μήνες. Εμείς ως βουλευτές έχουμε παραπάνω από δύο χρόνια ακόμα μπροστά μας. Μου φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρον όταν είπατε ότι είσαστε υπέρ του πρασινίσματος, φαίνεται να διαμορφώνεται συνένεση, αλλά φαίνεται πως οι ερμηνείες είναι πολύ διαφορετικές. Και μου φάνηκε ενδιαφέρον επίσης ότι είπατε ότι είσαστε ταυτόχρονα υπέρ των εξαγωγών. Αυτό ίσω οι εξαγωγέ δηλαδή για τη Δανία να παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά δεν συμβαίνει και παντού ότι όλη η παραγωγή δηλαδή κατευθύνεται στις εξαγωγέ σε όλε τι χώρε, Στην ατζέντα σα θα είναι σωστό να λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικέ εισαγωγέ και ότι οι εισαγωγέ εξακολουθούν και είναι μεγαλύτερε από τι εξαγωγέ. και ότι 30 εκατομμύρια εκτάρια χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια ζωοτροφών. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, διότι ορισμένα πράγματα έχουν ξεφύγει και δεν είναι λογικά και έχουν ξεφύγει λίγο από τον κύκλο και αν θέλουμε να αποκαταστήσουμε τον κύκλο στη γεωργία πρέπει να τα επαναφέρουμε τα πράγματα αυτά μέσα σε κάποια πλαίσια. Μιλήσατε το θέμα της προστασίας των ζώων, εξακολουθεί το θέμα αυτό και είναι πάρα πολύ έντονα ενδιαφέρον για την κοινή γνώμη. Υπάρχουν όμως και σημαντικότατα προβλήματα εφαρμογής. Εγώ δεν λέω ότι κάθε λίγους μήνες θα πρέπει να κάνουμε νέες προτάσεις στο Συμβούλιο δηλαδή. Θα πρέπει ωστόσο να εφαρμόσουμε με συνέπεια αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν. Και υπάρχει έλλειμμα εφαρμογής, όχι μόνο στις κότες και τα κοτόπουλα, αλλά υπάρχουν και άλλοι κανονισμοί που δεν εφαρμόζονται. Και πολλοί πολίτες και οργανώσεις πολιτών είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένοι από το λόγο αυτό. Χαίρομαι που θέλετε να βάλετε στην ατζέντα σας ένα θέμα το οποίο συζητιέται και στην ε, ε, κοινή γνώμη, δηλαδή η αντίσταση στα αντιβιωτικά. 25.000 νεκροί στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον χρόνο λόγω μικροβίων που ανθίστανται στα αντιβιωτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και στα πλαίσια της γεωργίας, γιατί έχει σχέση με τη γεωργία, έχει σχέση με την κτηνοτροφία. Μελέτε που έγιναν στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία έδειξε ότι κοτόπουλα 70% των κοτόπουλων σε αυτές τις 35 ημέρες που χάσαμε δυστυχώς το μικρόφωνο του μιλητή. Τώρα άναψε πάλι, αλλά δεν το είχε καταλάβει ο μιλητής. Στι 35 μέρες που ζουν τα κοτόπουλα λοιπόν, 70% από τα κοτόπουλα αυτά ε, καταπίνουν αντιβιωτικά. Το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί για τα πράγματα αυτά. Υπάρχει ανάγκη τη ανάληψη δράσης. Όλο και πιο βιομηχανική γίνεται η εκτινοτροφία και αυτό πρέπει να περιληφθεί ως θέμα σημαντικό κριτικής μέσα στην ατζέντα. Μιλήσαμε και για την κατασπατάληση των τροφίμων. Και είπαμε ότι μια από τις επόμενες χρονιές θα είναι το έτος κατά της κατασπατάλησης. Ε, πώς λοιπόν όμως τώρα η Γεωργία θα αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, ξέροντας όμως από την άλλη μεριά ένα 15 με 20% των τροφίμων πετιούνται τελικά στα σκουπίδια. Και αυτό πρέπει να παραμείνει μέσα στην εστίασή σας, ελπίζω και της δικής σας Προεδρίας. Κάτι που με εξέπληξε στη συζήτηση που έγινε στο μεσημεριανό γεύμα είναι που είπατε ότι ναι, πρέπει να κάνουμε το πρασίνισμα σε ορισμένες περιφέρειες. Αυτό είναι απαραίτητο και σίγουρα είναι και δυνατό, ώστε από την άλλη μεριά να μπορούμε να κάνουμε πιο εντατικέ τι καλλιέργειε. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Διότι θα σήμαινε, ο Άλμπερντές δεν με ακούει, αλλά Άλμπερντές θα σήμαινε, καλά, να κάνουμε αγρανάπαυση σε ολόκληρη τη Βαβαρία για να μπορούμε να κάνουμε εντατική καλλιέργεια στη Δανία. Δεν μπορεί να είναι αυτό ο στόχο των μέτρων μεταρρύθμισης. Σας ευχαριστώ. Γιατί οι προτάσεις της μεταρρύθμισης προβλέπουν μια οικολογικοποίηση, ας πούμε έτσι, σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Όχι να γίνει πιο οικολογική μία περιφέρεια ώστε να γίνει πιο εντατική η καλλιέργεια σε μια άλλη. Τις μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει να τις κρατήσουμε εστιασμένες ώστε να υπάρξει μια ισορροπία σε όλες τις περιφέρειες. Όχι να πούμε, όπως είπα, ορισμένοι είναι καλοί, ας γίνουν καλύτεροι και οι άλλοι να έχουν ελεύθερο για επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα των μέτρων του πρασινίσματος. Νομίζω λοιπόν έχουμε πολλή συζήτηση μπροστά μας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο Άγνιου κλείνει από τους συντονιστές. Thank you very much. Good afternoon, Minister. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα σας εκπλήξει να αρχίσω να μιλώ για αυγά. Και ίσως κάποιος σας πει, κύριε έχει τελικά ένα αυγό στο μετωπό σας, γιατί εδώ και 18 μήνες αυτό μας λέτε οι Βρετανοί. Πρέπει να σας πω ότι ακόμη υπάρχει μεγάλο ποσοστό μη συμμόρφωσης με το θέμα της συστοιχίας κλοβών. Θα μου πείτε γιατί. Διότι το σύστημα ήταν εντελούσιο καταρχάς, αλλά πρέπει να πω ότι υπήρχε στο τέλος και μεγάλος συμφόρηση, διότι έπρεπε πριν από τα Χριστούγεννα όλα αυτά τα πτηνά να τα βοηθήσουμε να βρούμε λύση. Πρέπει να πω ότι σε 10 μέρες ε, εξαιτία του προβλήματος που πρόκειται, διότι θα έλεγε η προθεσμία, μειώθηκε σε 50% αριθμός των πτηνών που δεν μπορούσαν, δεν θα συμμορφώνονταν με αυτό το, με το σύστημα. Τώρα συνέβη το ίδιο με τους Τσέχους. Στην Μεγάλη Βρετανία είπε ο υπουργό μας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή κυκλοφορούν αυγά με τέτοιου είδους ε, συνθήκες, διότι αυτό θα σημαίνει ότι καταστρατηγούμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το κάνουν οι Τσέχοι που πλημμυρίζουν με τα δικά του αυγά τον κόσμο. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε όμως, εάν κάνουμε όλοι ε, ό,τι κάνουμε οι Τσέχοι, σιγά σιγά θα δημιουργηθείτε γενικότερο πρόβλημα με τα πίνα αυτά. Έχετε έξι, μη, έχετε μήνες μπροστά σας κυρία Υπουργέ και νομίζω ότι κάτι παρατηρήσατε να βγουν από αυτού του είδους τα ε, και ακόμη και το τελευταίο πτηνά στο τέλος ε, της δικής σας προεδρίας. Εγώ είμαι αγρότης και πρέπει να σας πω ότι είναι μια αρκετά τυπική, τυπικό ακρόκτημα ε, το δικό μας. Πρέπει να πω ότι στο δικό μου ε, ακρόκτημα είμαστε με, έχουμε συμμορφωθεί με την ε, κοινοτική νομοθεσία. Έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό 4% που δεν συμμορφώνεται με τον τρόπο με τον οποίο κάνει τη Γεωργία μας με την ε, δική, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 6% δεν είναι μεγάλο ποσοστό, αλλά θα πρέπει να εγκαταλείψω ε, αυτό το μικρό ποσοστό, διότι διαφορετικά θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί. Οι πολλαπλές εσοδιές, όπως λέγεται. Δηλαδή, εάν σε, σε μικρές αναλογίες πρέπει να έρχεται στο αγρόκτημά σας τουλάχιστον τρεις διαδοχικές ε, εσοδιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους μικρούς γεωργούς θα τους ε, πλήξει πολύ περισσότερο από ό,τι τους μεγάλους και φοβούμε ότι θα πρέπει να έχουν τα πράγματα. Αν πείσετε τον ε, κύριο Τσόλος, τον Επίτροπο, να αυξήσει τα ποσοστά σε πιο λογικά ποσοστά θα βοηθήσετε ε, πολύ τους μικρούς Γιώργους. Είπε κάτι για τους δικαιούχους ο κύριο, ο συνάδελφος. Εάν δεν κάνουμε σωστά τα πράγματα και δεν έχουμε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης δίκαιους κανόνες, πάρα πολλοί αγρότες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις γέες και κυρίως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πλήξει τους νέους γεωργούς. Μπορείτε να το σκεφτείτε για να βρείτε λύσεις, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμη 13 συνέλευσεις που ζήτησαν λόγο. κύριος η κυρία Κανιέτε, με συγχωρείτε πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα η Δανέζικη Προεδρία να επιτύχει. Και θα πρέπει να υλοποιήσετε τους στόχους σας, ώστε να ανταποκριθείτε, όπως είπα τις προκλήσεις που έχετε. Έχω μία ερώτηση, σας το εύχομαι για Έχω μία ερώτηση. Άκουσα πολλές φορές ότι ένας από τους στόχους της Ινδανική Προεδρίας, στα πλαίσια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό, είναι να επιτύχει μείωση των κονδυλίων τα οποία προβλέπεται να δοθούν στην ΚΑΠ. Και θέλω να σας ερωτήσω, κυρία Υπουργέ, εάν τα κονδύλια που προβλέπονται για την ΚΑΠ μειωθούν, θα είναι πιο εύκολο για την Προεδρία να επιτύχει άμεσες πληρωμές και να έχει καλύτερη και πιο δίκαια ε, αγροτική πολιτική. Στην ε, Λετωνία και δική μας η Γεωργία έχουν τα ίδια ερωτήματα και τα ίδια ερωτηματικά, όπως και οι υπόλοιποι Γεωργοί. Αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν πιο δίκαιες άμεσες πληρωμές περισσότερες και πιο δίκαιες από ό,τι σήμερα. Ο κύριος Ταραμπέλα Ευχαριστώ Πρόεδρε κυρία Υπουργέ. Πέρα από τις προτεραιότητες που αναφέρατε, είναι αυτή που ανέφερε ο συνάδελφος ε, για την πτητικότητα των τιμών ε, των γεωργικών προϊόντων. Ξέρω ότι έχουμε ένα ενιαίο ντοσιέ το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο μια σημαντικής έκθεσης. Η παραγωγή είναι πολλές φορές ο αδύναμος κρίκος της όλης διανομής τροφίμων διότι η διανομή είναι πολύ οργανωμένη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους παραγωγούς στρεβλώνοντας λιγουλάκι τον, τον κανόνα της... του ανταγωνισμού. Είστε έτοιμοι να κάνετε αυτή την υποχώρηση. Κατά τη γνώμη μου ο κίνδυνος της ε, πτυτικότητας των τιμών των βασικών ε, τροφίμων ε, δεν φύγεται όσο θα έπρεπε από το κείμενο της Επιτροπής το οποίο εμείς θα, πρέπει να αλλάξουμε. Υπάρχει η κερδοσκοπία στα βασικά τρόφιμα η οποία δεν έχει ακόμη παταχθεί μέχρι σήμερα. Θα ήθελα, όπως επίσης υπάρχει και το θέμα των ε, καλλιεργιών για τα εναλλακτικά καύσιμα που επηρεάζουν στις τιμές. Θα μπορούσαμε λοιπόν να κάνουμε κάτι ούτως ώστε να σταματήσουμε όλη αυτή την τρομερή αστάθεια στις ε, τιμές ε, που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους γεωργούς. Σε ευχαριστώ. Μάρκ, ο Τζανκάρλος Πρόεδρε, Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τη νέα Δανέζικη Προεδρία, ελπίζοντας ότι θα κάνει σοβαρά τη δουλειά του στο επόμενο εξάμεινο. Η Επιτροπή Γεωργίας πάντοτε διαπετώ από ένα πνεύμα συνεργασίας με τα, με, τα άλλα ενδιαφερόμενα όργανα. Θα έπρεπε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι. Συμφέρον μας είναι να μπορέσουμε να δώσουμε φωνή στα εκατομμύρια των γεωργών που με τη δουλειά τους γεμίζουν το τραπέζι των άλλων εκατομμυρίων, πόσων εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε μία από τις βασικότερες πολιτικές σε κοινοτικό επίπεδο. Δεν πρέπει να χάσουμε λοιπόν την ευκαιρία να γράψουμε ένα κείμενο το οποίο να καλύπτει την πολύπλευρη πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, συγκεκριμένη κυρίως, όπως καινοτόμα και άλλο. Θα πρέπει να προσθέσουμε και στόχους. Στόχους για να ορίσουμε και την ουσία της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία. Ευχαριστώ Τζαν Κάρλο, Ντόρφμαν και μετά η Ράτσα Γκαρσία Πέρες. Ευχαριστώ Κύριε Υπουργέ, δύο σχόλια για την μεταρρύθμιση και μετά για, την, για τον κανονισμό ποιότητας. Η κυρία Κανιέτε είπε ότι χρειαζόμαστε δίκαιη κατανομή των κονδυλίων της ΚΑΠ. Αυτό δεν ισχύει βέβαια μόνο σε σχέση με την κατανομή ανάμεσα στις χώρες μέλη, ισχύει και για την... Χρειάζεται δηλαδή μια δικαιότερη κατανομή και μέσα στην ίδια τη χώρα μέλος μεταξύ των εκμεταλλεύσεων. Για παράδειγμα, για την Ιταλία, τη δική μου χώρα, υπάρχουν 20 περιφέρειες από 51 ευρώ ανά εκτάριο σε μία περιφέρεια μέχρι 510 ευρώ ανά εκτάριο στην πιο πλούσια περιφέρεια, σε αυτήν δηλαδή που δίνει τα περισσότερα. Είναι το δεκαπλάσιο. Αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη συζήτηση αυτή. Το δεύτερο τώρα, το πρασίνισμα δηλαδή, το greening, έρχομαι σε αυτό που είπε ο κύριος Ντέσ προηγουμένως. Για το πρασίνισμα πρέπει να σκεφτούμε ξανά αν ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε το μοντέλο του δεύτερου πυλώνα. Υπάρχουν σήμερα χώρες μέλη, μεταξύ αυτών και η Δανία, που λέγουν ότι στο δεύτερο πυλώνα δεν έγινε τίποτα και υπάρχουν άλλες χώρες που δίνουν το 30 και 40% των κονδυλίων για το πρασίνισμα. Τώρα να μπουν αυτά όλα στον πρώτο πυλώνα και να επιβληθεί το πρόγραμμα του πρασινίσματος με το ζόρι βρίσκονται ότι δεν είναι σωστό. Πρέπει να βελτιωθεί ο δεύτερος πυλώνας. Ένα θέμα τώρα για τον κανονισμό για την ποιότητα, όπου είμαι σκιώδης εισηγητής. Εκεί είναι σημαντικό να κινηθεί το Συμβούλιο. Έχουμε κολλήσει τώρα στον τριμερή διάλογο. Χρειάζεται να ρυθμιστεί ένα σοβαρό θέμα, ο προγραμματισμός δηλαδή των παραγωγών μέσω των οργανώσεων παραγωγών. Εάν δεν επιτευθεί κάποια πρόοδος, δεν θα μπορέσει να γίνει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και θα χρειαστεί δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Μιλήσατε και για το μικρό ντοσιέ του κρασιού, όπου είμαι σύμφωνος, είμαι και εισηγητής για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προσπαθήσουμε να το προωθήσουμε το ταχύτερο δυνατό, όπως είπατε, αν είναι δυνατόν και σε πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ Χέρμπερ ή Ράτσε και μετά ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, θα θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας και την παρουσίαση στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι η ενέργεια που επιδεικνύεται για τη δουλειά που σας περιμένει αυτό το εξάμεινο θα μεταφραστεί σε αποτελέσματα που θα είναι ευνοϊκά για όλη την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Είμαι σίγουρη ότι με τη συνεργασία που θα έχετε με την Επιτροπή μας θα υλοποιηθούν οι στόχοι σας. Στα πλαίσια τώρα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, νομίζω θα μπορούσαμε να έχουμε μια ευρύτατη συζήτηση. Ο καθένας από, εμάς, από θα μπορούσε να θέσει όλα τα ερετήματα τα οποία θέτει και στις προηγούμενες ε, Προεδρίες και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα διάφορα θέματα. Απλώς θέλω να πω κάτι πολύ απλό, να σας ζητήσω στα πλαίσια των συζητήσεων και των εργασιών που θα γίνουν και τα έργα της Προεδρίας σας να λάβετε υπόψη σε ένα θέμα το οποίο νομίζω είναι πρωταρχική σημασία. Το θέμα της ποικιλομορφίας της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Η Ευρωπή, Ευρώπη αποτελείται από διαφορετικές πραγματικότητες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η γεωργία της Δανίας σίγουρα με την γεωργία της χώρας μου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας. Λάβετε υπόψη λοιπόν αυτή την ποικιλομορφία της γεωργίας στην Ευρώπη, για πολλά θέματα. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων, για το πρασίνισμα, για όλα τα θέματα που έχουμε επιτάπητος, θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτό το στοιχείο της ε, ποικιλότητα. Όπως επίσης είπε και ο κύριος Καπούγιας, σε σχέση με τα ε, θέματα τα δημοσιονομικά, πολλές φορές το θέσαμε, μιλάμε για νέες προκλήσεις τις περισσότερες τις συμμεριζόμαστε, αλλά συνειδητοποιούμε σε μία συζήτηση για τον προπολογισμό, εάν δεν μπορέσετε να έχετε τα χρήματα στη τσέπη, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν το θέμα των κονδυλιών. Τώρα, όσον αφορά το πακέτο ποιότητας, όπως είπε και ο συνάδελφος Ντόρπφμαν, νομίζω ότι τους τελευταίους μήνες εργαστήκαμε πάρα πολύ εντατικά με την προηγούμενη πολωνική Προεδρία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το ίδιο θα γίνει και με τη δική σας Προεδρία, με την οποία ήδη είχαμε τις πρώτες επαφές. Απλώς θέλω να σας πω ότι η δουλειά που έχει γίνει από αυτό το θέμα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σχεδόν έχουμε φτάσει σε συστήματα ε, ποιότητας για τη γεωργία, σε συμφωνία για το 80% του περιεχομένου. Υπάρχει μας ένα θέμα το οποίο είναι θεμελιώδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το έχουμε πει πολλές φορές. Υπάρχει το θέμα που αφορά τον έλεγχο των ε, παραγόμενων ε, όγκων. Παρακαλώ λοιπόν να γίνει η συζήτηση από αυτού του θέματος και να μπορέσουμε να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο γενικότερα πρώτα απ' όλα. Και μετά θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Τι μας χωρίζει, τι μας ενώνει, αλλά θα πρέπει να ανοίξει η συζήτηση πρώτα απ' όλα για αυτό το θέμα. Διότι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαφορετικά θα είναι πολύ σύμφωνο να καταλήξουμε συμφωνία, να μην πω αδύνατον και για την, σε επίπεδο πρώτη ανάγνωση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για αυτό το θέμα μεταξύ μα. Και τελικά, δεν θα μιλήσω για τις κότες, όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει η ευημερία των πουλερικών. Ο κύριος Ανιώ το έχει κάνει πολλές φορές. Με ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει επίση είναι και τα πρόβατα. Τι γίνεται. Μιλούμε για δύο παρεμφερείς οδηγίες όσον αφορά την πλήρωση κάποιων κριτηρίων και για την ε, ηλεκτρονική ταυτότητα, αν θέλετε, των ε, προβάτων έχουμε μιλήσει εδώ και πολύ ε, καιρό πριν, γιατί είναι ένα θέμα πρώτερο από αυτό των ε, πτηνών και θα πρέπει να δούμε πώς έχει το θέμα της συμμόρφωσης ε, στο θέμα αυτό, διότι κάποιες χώρες δεν έχουν κάνει τίποτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την παρουσία της εδώ. Απογοητεύτηκα λίγο που δεν άκουσα περισσότερες λεπτομέρειες στην παρουσίασή της. Στην παρούσα φάση συζητούμε στην Επιτροπή Γεωργίας για δυόμιση χρόνια βέβαια την κοινή αγροτική πολιτική. Έχουμε μιλήσει πολύ και βρισκόμαστε όπως είπα σε μια φάση όπου αναζητούμε περισσότερες κατευθύνσεις, περισσότερες ιδέες, περισσότερο ψαχνό αν μπορώ να το πω έτσι. Θα ήθελα παρόλα αυτά να έρθω σε λίγα από τα σχόλια που κάνατε. Μιλήσατε για απλοποιημένη πολιτική. Τους τελευταίους μήνες έχω συνομιλήσει με πολλούς αγρότες στην περιφέρειά μου, στη Βόρεια Ιρλανδία, που θεωρούν τις προτάσεις της Κομισιόν εξαιρετικά περίπλοκες θεωρούν ότι αυτές θα συνεπάγονται ακόμα περισσότερη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τους αγρότες. Θα θέλαμε να μάθουμε εάν οι ιδέες της Δανικής Προεδρίας για την απλοποίηση της αγροτικής πολιτικής. Μα δεν μπορούμε να μιλούμε σαν να είναι το Άγιο Δισκοπότηρο και που υπάρχει υποτίθεται κάπου το πιστεύουμε και δεν υλοποιούνται ποτέ. Μιλούμε για, μια, για ένα τομέα πολιτικής που κοντεύει να καταστραφεί από τη ρύθμιση. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε εάν όντως θα οδηγηθούμε σε απλοποίηση της ΚΑΠ. Πάλι για το πρασίνισμα. Μιλάτε για το πρασίνισμα σαν να είναι η κατεύθυνση του μέλλοντος. Θέλουμε να μάθουμε και οι γεωργοί μας θέλουν να μάθουν. Πιστεύετε ότι τα μέτρα του πρασινίσματος θα μπουν στον πυλώνα 1, στον πρώτο. Πιστεύετε ότι τα μέτρα του πρασινίσματος που θα υλοποιηθούν όντως θα βελτιώσουν το περιβάλλον ή όπως εγώ είπα χθε εδώ στην Επιτροπή θα είναι δύσκολα για τους αγρότες και στη Βόρεια Ελληνική που έχουμε μικρές εκμεταλλεύσεις θα έχουν πρόβλημα για παράδειγμα με την εναλλαγή καλλιεργιών διότι τα μέτρα είναι υπερβολικά λεπτομερή και δεν θα μπορούν να είναι υλοποιήσιμα. Θα θέλαν λοιπόν και εγώ και οι αγρότες μου να μάθουμε εάν η Δανική Προεδρία έχει κάποια ξεκάθαρα πράγματα να τους πει, γιατί η Κομισιόν δεν φαίνεται να μπορεί να τους πει ξεκάθαρα πράγματα. Τα θέματα είναι δύσκολα. Εμείς έχουμε πολλά βοσκοτόπια εκεί. Τι θα γίνει με αυτά. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να επιδιώκει η παραγωγή να ανοίξει αγορές για εξαγωγές. Αλλά θέλω να μάθω εάν η επιδίωξη σύναψης εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει εν τέλει να οδηγηθεί σε βάρος, να οδηγήσει σε βάρος, να αποβεί σε βάρος της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και γιατί μπαίνει η Γεωργία στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη σηκώσει τα χέρια ψηλά και έχει πει αναγνωρίζουμε ότι ιτηθήκαμε και ότι οι διεθνείς συμφωνίες θα, οδηγηθούν, θα, θα αποβούν σε βάρος τελικά της Γεωργίας. Έχουμε τις διάφορες οδηγίες, αλλά χρειαζόμαστε κάποια κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αισθανόμαστε τρόμο, αλλά δεν έχουμε κανένα που να μας δώσει κατευθύνσεις. Αυτά χρειαζόμαστε από εσάς. Η κυρία Ραντς Γκαρσία και μετά η κυρία Πόλσεν. Ε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και Ρία ε, Υπουργέ και μιλούμε για τις προτεραιότητες σα. Άκουσα ότι τα πιο σημαντικά θέματα για σας είναι η μερία των Ζών και το μέλλον της ΚΑΠ. Όσον αφορά την στρατηγική για την ευημερία των ζώων, θα θέλα τελικά να αφήσουμε τις ε, αηδίες και τις προκαταλήψεις και να, με επιστημονικά στοιχεία να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Διότι μέχρι τώρα αυτό το οποίο έκαναν η Επιτροπή και το Συμβούλιο είναι να βασίζονται ώρες-ώρες σε ανόητα επιχειρήματα και σε δυσυδαιμονίες για να κάνουν κάτι. Και νομίζω ότι ποτέ δεν βασίστηκαν σε επιστημονικά στοιχεία. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που αναφέρατε για την ΚΑΠ. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα αυτό. Με απασχολεί διότι είμαι από μία χώρα στην οποία το μέλλον της ΚΑΠ είναι κάτι στο οποίο, ε, το οποίο αφορά το μέλλον πάρα πολλών οικογενειών και την βιωσιμότητα πολλών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Γι' αυτό, μιλώντας για πρασίνισμα, θα πω το εξής αυτά τα οποία προβλέπει στις ε, προτάσεις της Επιτροπή δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε για τους ελαιώνες ούτε για την καλλιέργεια τους οριζόνες. Διότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ισπανία, στις οποίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν ε, οι αρχές που πρεσβεύει στην πρότασή της Επιτροπή. Θα πρέπει λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη αυτό που είπαμε για την ε, διαφοροποιήσεις και την ποικιλότητα, να των διαφόρων γεωρικών εκμεταλλεύσεων να γίνουν ε, να ακουστούν οι απόψεις όλων για να μπορέσει να γίνει μία σωστή πολιτική. Τώρα όσον αφορά την ε, τιμή του ελαιολάδου θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε την πολιτική διαμόρφωση των τιμών να την αναθεωρήσουμε διότι είναι πεπαλαιωμένη, βασίζεται σε αρχές που δεν ισχύουν πλέον και θα πρέπει κυρίως για την τιμή αναφοράς, ε, να κάνουμε ε, κάτι για να βοηθήσουμε τους ελαιοπαραγωγούς να προχωρήσουν. Διότι δεν μπορούν καν να προχωρήσουν σωστά αυτοί οι οποίοι δεν ε, είναι σε ένα συνεταιρισμό. Και εμείς θέλουμε ο καθένας από μόνος να μπορέσει να το κάνει. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει κάτι για να μην εκμεταλλεύονται το τομέα μόνο κάποιοι λίγοι παραγωγοί. Επίσης, στα πλαίσια της ε, εισήγησης που θα γίνει για τις ε, ε, περιφέρειες της ε, μακρινές, αν θέλετε, τις υπερπεριφερειακές, τι προβλέπετε να κάνετε. Μας ενδιαφέρει εμάς τα Κανάρια, μας ενδιαφέρει τι θα γίνει στα πλαίσια των, της Γαλλίας και της Πορτογαλίας. Κύριε Πούλσαν, κυρία Αντιπρόεδρε, σας καλωσορίζω. Όσον αφορά τα αντιβιωτικά, είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσαμε εκτενώς, δεν θα το αναφέρω. Παρά το γεγονό ότι είμαι συγγήτρια για το θέμα αυτό. Σε όλη αυτή τη συζήτηση αυτό το οποίο εμένα με ανησυχεί είναι η γραφειοκρατία. Φοβούμαι ότι θα έχουμε ένα σύστημα πιο πολύπλοκο από αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα σαφές, με σαφή νομοθεσία, ώστε να μπορούν οι πάντες να το καταλάβουν το σύστημά μας. Όχι ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται κείμενο θα καταλαβαίνουν μόνο κάποιοι βουλευτές και η γραμματεία τους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη φοβούμε λοιπόν τη γραφειοκρατία. Απ' την άλλη σκέφτομαι την ελευθερία που πρέπει να έχει κάθε γεωργός. Ώστε ο καθένας να μπορεί να βασίζεται στα εισοδήματά του. Πρέπει να βασιστούμε λοιπόν στις νέες ιδέες, στις νέες αντιλήψεις, στην καινοτομία και θα πρέπει να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να υποφεληθούν από αυτές τις καινοτόμες ιδέες. Θα πρέπει παντού λοιπόν στην Ευρώπη να μπορέσει ο καθένας να δοκιμάσει τις ιδέες του και να τις θέσει εφαρμογή για να δει αν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Διότι έχω την εντύπωση ότι σήμερα στην Ευρώπη ζούμε σε έναν κόσμο ε, κρίσης οικονομικής και δημοσιονομικής τρομερό και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γεωργούς. Γιατί πέστε μου, ποιοι είναι οι γεωργοί που μπορούν σήμερα να δανειστούν για να υλοποιήσουν ε, τις ε, ιδέες τους και τις αντιλήψεις τους και τις καινοτομίες που θέλουν να εισαγάγουν. Στη δεκαετία του 80 στην Σουηδία υπήρχαν κάποιες εγγύσεις και μπορούσαν οι γεωργοί κάτι να κάνουν. Θα μπορούσαν να πηγαίνουν ε, ε, στις τράπεζες και να ζητούν ειδικέ πιστώσεις για τέτοιου είδους θέματα. Θα κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει και σήμερα στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα. Ας το προσπαθήσουμε. Σε συνδυασμό με τι μπορούμε να κάνουμε επίσης και στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης. Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι το παρεμφερέ σήμερα. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα. Νομίζω, Φερρυπίν, ότι όσον αφορά το θέμα της προστασίας των ζώων, έχουμε επιστημονικές μαρτυρίες και στοιχεία που μας αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πάρα πολύ ασφαλή συστήματα ε, διατροφής των ζώων. Αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθά πάρα πολύ τους γεωργούς εάν ξέρουν κάτι τέτοιο, ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και είναι και μια εγγύηση για τη δημόσια υγεία. Και εγγύηση ότι παράγουμε ασφαλή προϊόντα. Βεβαίως, θα πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια, ώστε ό,τι κάνουμε να μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη, ώστε να κάνουμε πολιτικές αποδοτικές. Η γεωργία είναι θέμα ευθύνης όλων μας και για θέματα της ενεργειακής απόδοσης και για την βιωσιμότητα και για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να γίνει σε θέματα ενέργειας αυτάρκης η Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και αν χρησιμοποιήσουμε όλα τα οργανικά απόβλητα τα οποία έχουμε για να παράγουμε και βιοκαύσιμα, μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες οικονομίες και στον τομέα της ενέργειας. Και έτσι θα συνεισφέρει η γεωργία και στην μείωση των εκπομπών ε, μεθανίου και διοξιδίου τόσο από την παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε να είναι έτσι η γεωργία μας αύριο. Τώρα, ίσως είμαι λίγο εκτός θέματος για θέματα διότι μιλούμε εδώ για μεταρρύθμιση της ΚΑΤ. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να σκεφτούμε το μέλλον με κάποια φαντασία και με ελευθερία, ώστε να μπορέσει ο καθένας να εκφράσει τις ιδέες του. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε Πόλσον, κύριε Ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα μαζί σας, στην αρχή της Προεδρίας σας, το πρόγραμμά σας, το πρόγραμμα εργασιών σας είναι τεράστιο και μόνο διαβάζοντας τους στόχους σας ανησυχώ και περισσότερο ότι πηγαίνουμε προς μια Ευρώπη πολλαπλών, πολλαπλών ταχυτήτων και στον αγροτικό τομέα και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή οδηγιών και σε ό,τι αφορά την εφαρμογή κανονισμών. Και αυτό θα, θα, προτελέσει, θα αποτελέσει πρόβλημα για τον ανταγωνισμό, διότι αν υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή των κανονισμών, είτε πρόκειται για τις συστοιχίες κλοβών ορνήθων, είτε πρόκειται για άλλα θέματα, μπαίνουμε εμείς μόνοι μας σε προβλήματα, γιατί αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν τους κανονισμούς τελικά προχωρούν μπροστά ταχύτερα. Και αυτό ισχύει και για την προστασία των ζώων. Και δεν παραμένουμε μέσα σε πλαίσια προτύπων. Θα έχουμε τα σημαντικά προβλήματα διότι οι αγρότες εκείνοι οι οποίοι καταφέρουν τελικά να προσαρμοστούν θα αντιμετωπίσουν εν τέλει μειονεκτήματα ανταγωνισμού. Θα είναι μειονεκτικά ε, ανταγωνιστικοί διότι όλα αυτά έχουν, η προσαρμογή δηλαδή στους νέους κανονισμούς συνεπάγεται κόστος. Εφόσον όμως ο αγρότης επενδύει για να ε, σεβαστεί τους κανονισμούς πρέπει να έχει και κάποιο πλεονέκτημα. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν μήπως η καινοτομία και η πρόοδος εν τέλει αποτελέσει κίνδυνο, απειλή για την Ευρώπη. Εάν δεν προχωρήσουμε όμως, πώς θα συνεχίσουμε να παίζουμε πρωτοπόρο ρόλο στην παγκόσμια αγορά, όταν πολλές άλλες χώρες θα μας ξεπεράσουν. Και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, το αυτό ούτε ως Ευρωπαϊκή Γεωργία. Και εξετάζοντας όλο αυτό το πακέτο πρέπει να δούμε πού θα, πώς θα προχωρήσουμε τώρα με το προπολογισμό και με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εν ώψη και της οικονομικής κρίσης, πώς είναι δυνατόν να σχεδιάσουμε το μέλλον της Γεωργίας όταν γνωρίζουμε καν ποια δημοσιονομική βάση θα έχουμε, πόσα χρήματα θα έχουμε. Είναι ζήτημα εφαρμοσιμότητας. Χρειαζόμαστε πρώτα ένα πλαίσιο δημοσιονομικό για να μπορούμε να ξέρουμε και να αποφασίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα τεράστιο ευχολόγιο για το ποια πράγματα θέλουμε να κάνουμε και τελικά να αποδειχθεί ότι δεν έχουμε λεφτά. Και ναι, οι χώρε μέλη έχουν το δικαίωμα να χρώνονται, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει. Δεν μπορεί να, να δανειστεί. Πώ λοιπόν θα τα εφαρμόσουμε αυτά τα πράγματα, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε πρόοδο και στο δημοσιονομικό τομέα για να ξέρουμε προς τα πού βαδίζουμε. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι και το greening. Λέτε καθαρά ότι εσείς θέλετε περισσότερη ευελιξία. Δεν θέλετε αύξηση της γραφειοκρατίας. Αν δεν θέλετε αύξηση γραφειοκρατίας, αν θέλετε περισσότερη ευελιξία, τότε από τη σκοπιά της Δανίας ίσως πρέπει να σκεφτείτε ότι το greening, το πρασίνισμα πρέπει να περάσει περισσότερο στον δεύτερο πυλώνα, που είναι ευκολότερο να υπάρξει αυτή η ευκαμψία. Όπω έχουμε πει κατά επανάληψη εδώ, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ διαφορετική. Οι αφετηρίε των διαφόρων γεωργικών οικονομιών στι χώρε μέλη είναι πολύ διαφορετικέ. Εξετάστε και τι νέε χώρε μέλη που βρίσκονται σε πολύ διαφορετική φάση ανάπτυξη από τι παλαιότερε. Το ίδιο σημαντικέ διαφορέ υπάρχουν μεταξύ βορρά και νότου. Βρίσκω λοιπόν ότι είναι σχεδόν άνευ λύσος το πρόβλημα εάν δεν τα θεμελιώσουμε αυτά όλα, τις προσπάθειες αυτές όλες νομικά. Και η ανακατανομή, το καταλαβαίνω αυτό θέλετε να κάνετε μεταξύ παλαιών και νέων χωρών μελών. Και οι χώρες μέλη όπου δεν έχουν κάνει ακόμα την προσαρμογή πρέπει να προσαρμοστούν. Εγώ αναμένω και από την πλευρά του Συμβουλίου να βάλετε τις κατευθύνσεις για την πορεία αυτή. Γιατί αν θέλουμε μέχρι το 2020 να τα έχουμε επιτύχει αυτά, τις προσαρμογές αυτές, πρέπει να βάλουμε την πορεία από τώρα. Και στη Γερμανία κάναμε τεράστια προσπάθεια για την προσαρμογή. Και μόνο με τον προγραμματισμό και τη σκληρή δουλειά μπορέσαμε να το πετύχουμε. Δεν σας ζηλεύω λοιπόν για αυτά που έχετε να αντιμετωπίσετε. E Ευχαριστώ Μπρίτα. Η κυρία Σέντεμολς και μετά ο κύριος Γιάρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί Μέτε, καλώς όρισες. Καλώς όρισες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λες ότι πράγματι για έξι μήνες οι βοηθοί σου πρέπει να εργαστούν σκληρά και εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου όταν βλέπω το πρόγραμμά σου, το οποίο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο. Είναι απαραίτητο να έχουμε ένα φιλόδοξο πρόβλημα, ε, πρόγραμμα σχετικά. Είναι καλό να έχουμε ένα πρόγραμμα ε, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μια βιώσιμη ΚΑΠ. Θα ήθελα να μιλήσουμε για την σπατάλη των τροφίμων. Συμφωνείτε? Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε ότι έπρεπε να μειώσουμε σημαντικά το ποσοστό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τα αντιβιωτικά και η, αντίσταση στα η αντοχή στα αντιβιωτικά. Η Προεδρία θα μπορούσε να εισάγει μία απαγόρευση πώλησης φαρμάκων για να χρησιμοποιούμε καλύτερα τα αντιβιωτικά στον κτηνιατρικό τομέα. Τι σκέφτεσαι γι' αυτό. Επίσης, τρίτον, πολλοί το σκέφτονται από τους συναδέλφους και είναι πρόβλημα για πολλούς διαπιστώνουμε σχετικά με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων στον τομέα της γεωργίας, της προστασίας των ζώων, οι χώρες δεν προχωρούν όλες με την ίδια ταχύτητα. Συζητήσατε για αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε στο μέλλον όλοι μαζί να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα και πιο συγκεκριμένα αυτούς τους κανόνες. Αυτό είναι αποφασιστικό για τους γεωργούς. Χρειάζεται να έχουμε ίδιο ανταγωνισμό για όλους σε ορισμένες ε, χώρες οι νομοθεσίες εφαρμόζονται και όχι αλλού. Τι θα κάνει η Δανία για να λύσει το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ που ήρθες και σε ευχαριστώ που υποσχέθηκες έναν θετικό διάλογο με το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Η φάση στην οποία εισερχόμαστε είναι σημαντική. Ελπίζω ότι με κοινή προσπάθεια δική σας και δική μας θα μπορέσουμε να προωθήσουμε λίγο την κοινή αγροτική πολιτική και μάλιστα με επιτυχία. Τέσσερα σύντομα σχόλια ή ερωτήσεις όπως θέλετε. Πρώτη ερώτηση. Πότε νομίζετε ότι θα γνωρίζουμε περίπου πόσα χρήματα θα έχουμε στη διάθεσή μας το κάτω της γραφής εκπροσωπείται μια χώρα μέλος και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι μπορούμε να αναμένουμε για το μελλοντικό σχεδιασμό ως κονδύλια δηλαδή. Εγώ χάρηκα που είπατε ότι αγωνίζεστε κι εσείς υπέρ της απλούστευσης και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Η δική μου παράκληση είναι μη λησμονήστε τα λόγια σας αυτά ποτέ. Σε κάθε λεπτομέρεια Κάθε λεπτομέρεια που θα εγκρίνουμε εδώ θα πρέπει να οδηγεί στη μείωση γραφειοκρατίας. Να μην λησμονείτε και την εναρμόνιση. Άλλοι συνάδελφοί μου προηγουμένως τόνισαν πόσες πολλές διαφορές υπάρχουν κάτω από αυτή την κοινή στέγη της κοινή αγροτικής πολιτικής. Ωραία είναι η επικεφαλίδα, η αγροτική πολιτική, αλλά από κάτω υπάρχουν δεκάδες διαφορές από τις άμεσες πληρωμές μέχρι το επίπεδο εφαρμογής των διατάξεων. Ε, ε, δεν έχει τελειώσει μια μεταρρύθμιση και αρχίζει η επόμενη. Αυτό βέβαια δεν δημιουργεί εμπιστοσύνη στους αγρότες. Μια παράκληση ακόμη για την προστασία των ζώων και τα προβλήματα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Κανονικά φέτος θα πρέπει να απαγορευτούν οι συστοιχίες κλοβών ορνήθων. Γνωρίζουμε ότι 12 χώρες μέλη ακόμα δεν τα έχουν καταφέρει που πάει να πει περίπου 30% της παραγωγής αυγών γίνεται από κότες που δεν θα, με τρόπο που δεν επιτρέπεται. Δηλαδή στην πραγματικότητα είναι απαγορευμένη η παραγωγή αυτή. Ανεξαρτήτως του ότι αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, δείχνει πόσο μειωμένη και αξιοπιστία της πολιτικής. Δηλαδή φτιάχνουμε διαρκώς οδηγίες και κανονισμούς και δεν καταφέρνουμε ένα κανονισμό που είχε 12 χρόνια μεταβατική περίοδο. Εγκρίθηκε πριν από 12 χρόνια και δεν καταφέραμε ωστόσο ακόμα να τον εφαρμόσουμε. Η ερώτησή μου είναι πώς θα συμβάλλεται να αποκατασταθεί ο ισότιμος ανταγωνισμός και ανάμεσα στους κτηνοτρόφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πέτε, η Ελίζαμπεθ. Και μετά ο Σπύρος Δανέλης για να τελειώνουμε. Ευχαριστώ κύριε... κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Διαρωτώ με τι εντυπώσεις θα πάρετε μαζί σας όταν θα εγκαταλείψετε την αίθουσά μας και πώς θα μπορέσετε κάπως να διαρθρώσετε στο μυαλό σας αυτές ε, τις απαιτήσεις που προβάλαμε. Εγώ σημείωσα ότι είπατε ότι είστε υπέρ της βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης. Εγώ διαρωτώ με αυτή η πράσινη ανάπτυξη πώς διαμορφώνεται και στην χώρα σας, στη Δανία. Πώς την εφαρμόζετε. Άλλωστε αυτή τη χώρα εκπροσωπείτε. Ακούσατε πόσο πολύ μας απασχολεί το θέμα το πρασίνισμα στον πρώτο πυλώνα, άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στο δεύτερο πυλώνα, πώς το σκέφτεστε. Μιλήσατε για την ασφάλεια τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών. Αναφερθήκατε και στην αντίσταση στα αντιβιωτικά. Σημαντικό θέμα και εδώ λοιπόν έχω συγκεκριμένο ερώτημα. Τι σκέπτεστε να κάνετε και ιδίω υπό τον τίτλο «Προστασία του καταναλωτού» Πώς δηλαδή θα μειωθεί η επιρροή των αντιβιωτικών στον άνθρωπο. Δηλαδή πώς θα αποφύγουμε αυτή την ε, ενίσχυση των ε, μικροβίων. Και για την προστασία των ζώων ακούσατε από πολλούς συναδέλφους πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν για την προστασία των ζώων και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ειδικότερα μέσα στην αγροτική πολιτική. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα της προστασίας των ζώων εγώ είμαι αρμοδία του Λαϊκού Κόμματος για την προστασία των ζώων και έχω κάνει και την πρώτη έκθεση το 2006. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Πάουλσεν για τα όσα είπε. Και γι' αυτό δεν θα επανέλθω. Σας επισημαίνω όμως με το κανονισμό για τις κότες, με το κανονισμό για τα χοιρινά. Οι φορολογούμενοι, και ακούσατε πολύ συχνά να σας ρωτάμε για τον προϋπολογισμό, ο φορολογούμενος λοιπόν μας κατηγορεί ότι το τμήμα αυτό, δηλαδή η μη εφαρμογή των κανονισμών, ο φορολογούμενος την θεωρεί μεγάλη αποτυχία της, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να φτιάχνουμε καινούργια νομοθετήματα, αλλά πώς θα προχωρούμε όταν δεν εφαρμόζονται τα παλιά. Αυτό πώς θα το περιλάβετε στο νέο πρόγραμμα εργασιών. Και θα ήθελα επίσης να ακούσω από εσά μετά από την συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορούμε να περάσουμε και πέραν αυτής, αυτού του πλαισίου προστασίας των ζώων. Δηλαδή να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Με, ποιο, με ποια κατεύθυνση, με ποιο δρόμο. Ευχαριστώ Ελίζαβε. Ο Σπύρος Νανέλης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλή δύναμη και καλή δουλειά και αποτελεσματική επίσης. Ε, ζήτησα το λόγο για να θέσω ένα διαφορετικό θέμα που δεν ακούστηκε. Ε, κατά την γνώμη μου υψηλής ε, και συμβολικής αλλά και ουσιαστικής αξίας. Και αναφέρομαι στην αναγκαιότητα ουσιαστικής στήριξης της βιοπικιλότητας και κυρίως των παραδοσιακών ευρωπαϊκών σπόρων. Όπως επίσης και την ανάγκη σύνδεσής τους με την ε, πολιτισμική κληρονομιά των χωρών μελών και της ίδιας της Ένωσης. Ε, ξέρετε, με ενοχλεί πάρα πολύ μια ιδέα που με βασανίζει καιρό τώρα, ότι η γενιά η δική μας έχει το θλιβερό προνόμιο μιας πολύ μεγάλης ε, ιστορικής ήττας, απώλειας. Πριν από 10.000 χρόνια περίπου, ε, το είδος μας, ο Homo sapiens, πέρασε από την παλαιολιθική εποχή στη νεολιθική, ε, ελέγχοντας το σπόρο, ελέγχοντας την παραγωγή των προϊόντων των αγροτικών και εξημερώντας κάποιες φυλές ζώων. Ε, η δική μας γενιά έχασε τον έλεγχο αυτό, αφιόμενη στην ευκολία του έτοιμου παραγωγικού υλικού, το οποίο ελέγχει ένα πολύ μικρό παγκόσμια ολιγοπόλιο, ε, παράγοντας υβριδικά, υβριδικούς σπόρους, ε, ελέγχει αυτό το λιγοπόλιο και την παραγωγή. Ο παραγωγός δεν μπορεί να παρέμβει στη σπορά του, δεν ελέγχει την παραγωγή του και έτσι ε, τα παιδιά μας δεν τρών δεν μπορούν να φάνε και δεν μπορούν να γευτούν απλά αγροδιατροφικά προϊόντα που εμείς προλάβαμε, όπως είναι η ντομάτα, όπως είναι το αγκούρι, όπως είναι πάρα πολλά χυπευτικά. έτσι νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα πολύ μεγάλης σημασίας το οποίο μας διαφεύγει. Ε, σκέφτεστε ότι η δική σας Προεδρία θα μπορούσε να βάλει τα πρώτα βήματα για την ίδρυση ας πούμε ε, ενός μιας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Σπόρων και κάνοντας ουσιαστικές κινήσεις για την ε, προστασία και τη διαιώνιση των σπόρων που, του, του παραδοσιακού πολλαπλασιαστικού υλικού του ευρωπαϊκού που απειλείται με εξαφάνιση. Ευχαριστώ. Eh, ευχαριστώ Σπύρο, ευχαριστώ όλους. Όπως βλέπεις αγαπητοί Μέτε, 19 συνάδελφοι μίλησαν παρότι η συζήτηση ήταν εκτενής ε, δηλαδή στο Συμβούλιο είστε 27. Έχεις το λόγο τώρα για να απαντήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι όλοι θέλετε να λάβετε το λόγο γιατί τα θέματα είναι πολύ σημαντικά και όλοι και όλες θέσατε σημαντικά θέματα προς συζήτηση και είμαι βεβαία ότι μπορούμε να συζητήσουμε για πολύ καιρό τα πράγματα αυτά διότι χρειάζεται να βρούμε λύσεις στα προβλήματα αυτά και που ανέφερα εγώ και που αναφέρατε εσείς και μάλιστα κοινέ λύσεις αλλά νομίζω ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητήσουμε νέες λύσεις. Λύσεις που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Δεν χρειαζόμαστε χθες νέες λύσεις, χρειαζόμαστε νέες λύσεις. Αυτά θα συζητήσουμε πού νομίζουμε ότι πηγαίνουμε, πού νομίζουμε ότι πηγαίνει ο κόσμος. Πρέπει να αντιληφθούμε και για ορισμένους από εσά, μάλλον θα πω κάτι το προσωπικό αλλά πιο μετά. Θυμηθείτε τώρα ότι εγώ είμαι προεδρία, δεν είμαι Δανέζα Υπουργό, βεβαίω και είμαι Δανέζα Υπουργό, αλλά δεν είμαι τώρα εδώ Δανέζα Υπουργό. Μη μου ζητείτε λοιπόν να πάω στις Βρυξέλλες, έτσι τους είπα, και να γυρίσω πίσω να σας φέρω όλα αυτά τα πράγματα που, που θέλετε εσείς για τη Δανία. Έτσι είπα στους δικούς μου. Είμαι υποχρεωμένη να αναζητήσω κοινό έδαφος και όχι να φέρω τα δικά μας μικρότερα θέματα. Βέβαια μερικοί Δανείοι ψηφοφόροι μου δεν συμφωνούν, αλλά η δική μου φιλοδοξία είναι αυτό ακριβώς να κάνω. Θα απαντήσω λοιπόν στις ερωτήσεις σας για τη Δανία, αλλά δεν θα αποδώσω εκεί την μεγαλύτερη σημασία, διότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο και σε αυτόν πρέπει να προσαρμοστούμε. Ναι, έχουμε εισαγωγές. Έχουμε όμως και εξαγωγές. Και πολλές από τις εξαγωγές μας βασίζονται στις εισαγωγές. Και το αντίθετο. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται να εξετάσουμε είναι τι μπορούμε να κάνουμε Τι μπορούμε να προσφέρουμε δηλαδή σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, το οποίο να επιζήσει. Τι μπορούμε να προσφέρουμε εμείς. Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Οι οικονομολόγοι του ΩΣΑ συμφωνούν μαζί μου, ή εγώ συμφωνώ μαζί τους βέβαια, νομίζω ότι μάλλον αυτοί τα σκέφτηκαν πρώτοι αυτοί, ότι η πράσινη οικονομία θα παραμείνει μαζί μας. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην ε, παγκόσμια αγορά στη βάση χαμηλών μισθών. Αυτό δεν γίνεται, αλλά μπορούμε να ανταγωνιστούμε στην βάση της υψηλής ποιότητας, της υψηλού επίπεδου προστασίας των ζώων, της καινοτομίας, δηλαδή νέων προϊόντων. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Και βέβαια, χρειαζόμαστε βιώσιμες οικονομίες με μικρή παραγωγή, μικρή, οι μικρές περιφερειακές μονάδες. Μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό κάτι που πολλοί και πολλές από σας είπατε ότι χρειάζεται ίση εφαρμογή σε όλες τις χώρες μέλη. Η ισοδίκαιη κατανομή, δηλαδή η ισοδίκαιη εφαρμογή για παράδειγμα για την προστασία των ζώων ισχύει αυτό. Και συμφωνώ. Μιλήσαμε και για τις οτόκες όρνηθες στο Συμβούλιο, μιλήσαμε και για τις ε, χειρομητέρες που ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου του 2013 και ζητήσαμε από την Κομισιόν να είναι ιδιαίτερα αυστηροί, σκληροί με τις χώρες μέλη. Μας είπαν πότε, χθες, σήμερα, χθες το απόγευμα, ότι έχουν αρχίσει διαδικασίες προσφυγής επί παραβιάση κατά 14 χωρών για την εφαρμογή του κανονισμού για τις οτόκες όρνηθες που πάνε να πει ότι αντέδρασαν γρήγορα. Είμαστε στο Γενάρη και έχουν ήδη αρχίσει τις νομικές διαδικασίες. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πολίτες που ζητούν προστασία των ζώων. Έχουμε ένα κοινοβούλιο που θέλει ισοδίκαιη εφαρμογή σε όλες τις χώρες και το Συμβούλιο το ίδιο. Όμως μια από τις μελλοντικέ απαντήσεις είναι όταν θα ψηφίσουμε κανονισμούς μακροπρόθεσμα 12 χρόνια. 12 χρόνια είχαμε μεταβατική περίοδο για να εφαρμοστεί ο κανονισμός αυτός αυτό τόσο μακρές περιόδους δίνουμε γιατί δεν θέλουμε η παραγωγή να διακοπεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Να τους δώσουμε λοιπόν μεγάλη μεταβατική περίοδο για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον για την προστασία των ζώων είναι να βάλουμε διάμεσους σταθμούς έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα προχωρεί στις χώρες. Γιατί συμφωνώ απόλυτο ότι είναι απολύτως απαράδεκτο να έχουμε αγρότες που να ανταγωνίζονται από χώρα σε χώρα αλλά και μέσα στις ίδιες χώρες με διαφορετικούς όρους. Χρειαζόμαστε λοιπόν ισότιμο ανταγωνισμό και στα πλαίσια της προστασίας των ζώων. Αυτό λοιπόν είναι βέβαια ένα σημαντικό θέμα. Το ίδιο σημαντικό είναι να πούμε θα κάνουμε μια διάσκεψη για την προστασία των ζώων και θα εξετάσουμε ορισμένε από τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, την, για δείκτες της προστασίας των ζώων. Αυτό ίσω είναι ένας νέος εξέταση του θέματος. Να μην έχουμε αυτόν τον αυστηρό κανονισμό που προκαλεί η γραφειοκρατία κτλ. Ίσως μερικά από τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν εφόσον οι καταναλωτές το ζητούν, αλλά και με δείκτες. Γνωρίζουμε ότι γίνονται αυτά. Ξέρω ότι υπάρχουν δανείοι χειροτρόφοι που παράγουν χείριο κρέας για βρετανικά για σούπερ μάρκετ. Και αυτό είναι καλό γιατί έχουν ένα έξτρα κίνητρο, έχουν παραπάνω λεφτά. Αυτά είναι πράγματα που θέλω να συζητήσω. Και να βασιστούν σε επιστημονική θεμελίωση. Ας γυρίσω λίγο πίσω να πω αυτό το προσωπικό πράγμα. Εγώ μεγάλωσα στην Ήπεθρο και σπούδασα αγρονόμος. Και εργάστηκα πριν να περάσω στο Υπουργείο Προστασίας του Καταναλωτού και έγινα και βουλευτής. Δηλαδή μια ζωή στην αγροτική παραγωγή. Και πιστεύω ακράδαντα ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες έχουν την ικανότητα να προχωρήσουν. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι αγρότες θα μπορέσουν να συνεισφέρουν στις κοινωνίες μας. Ακόμα και σε περίοδο κρίσης και χρειάζεται να τους βοηθήσουμε ώστε να μην κάνουν αυτά που κάνανε χθε, αλλά αυτά που τους ζητούμε να κάνουν αύριο. Αυτό είναι δική μου προσωπική λοιπόν άποψη με το ιστορικό που έχω. Πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον για τους αγρότες, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε. Καμιά φορά λέω στους δανούς αγρότες, αλλά μην τους το πείτε, ότι χρειάζονται λίγο σπρόξιμο. Αλλά βοηθάει αυτό. Επανέρχομαι τώρα στην Προεδρία. Όταν θα έρθουμε στις συγκεκριμένες συστάσεις και προτάσεις, πυλώνας 1 ή 2, θα το συζητήσουμε το Μάρτιο. Αυτό που είναι σημαντικό να πούμε είναι όταν θα συζητήσουμε την ανακατανομή να μην συζητήσουμε μόνο για τον πυλώνα 1 πρέπει να περιλάβουμε και τον δεύτερο πυλώνα. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα είναι σημαντική. Το ίδιο συζήτηση για το πρασίνισμα. Πολλοί λένε ότι υπάρχουν προβλήματα με το greening στον πρώτο πυλώνα. Είναι μία πρόταση. Η πρόταση θα μπορούσε να είναι να επεκταθεί το μενού του πρασινίσματος στον πρώτο πυλώνα, ώστε να υπάρχουν περισσότερες επιλογές, περισσότερες δυνατότητες για την ανάπτυξη του πρασινίσματος. Η δυσκολία εδώ είναι η Ευρώπη των 27 στην Ευρώπη των 27 είναι να βρεθούν τα ίδια στοιχεία πρασινίσματος για 27 χώρες μέλη με διαφορετικά εδάφη, διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικό κλίμα, ακόμα και διαφορετικές γλώσσες. Όλα είναι διαφορετικά. Και όμως παρόλα αυτά είμαστε, εξακολουθούμε και είμαστε ενωμένοι. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι αναζήτηση κοινού εδάφους. Δηλαδή ίσως χρειαζόμαστε περισσότερες δυνατότητες πρασινίσματος, να έχει κανείς δηλαδή ένα μενού να μπορεί να επιλέγει. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα ως Προεδρία είναι ότι αυτό δεν θα πρέπει να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, το πρασίνισμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, αυτές είναι ορισμένε από τις συζητήσεις που θα διεξαγάγουμε. Για παράδειγμα, επίσης, η κατανομή μεταξύ των χωρών μελών. Και ορισμένοι εξημών, αγαπητά μέλη, μιλήσατε για την εσωτερική κατανομή μέσα σε κάθε χώρα μέλος. Αυτό είναι δύσκολο θέμα. Σα το ομολογώ, διότι αυτό το κρίνουν οι ίδιες χώρε μέλη. Ή το έκαναν στην, ιστορικά. Κάθε χώρα μέλος απεφάσιζε δηλαδή μόνη τη. Αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Αυτό πιστεύω. Και βρίσκω ότι βλέπω ότι ο πρόεδρος συμφωνεί μαζί μου. Δόξα τω Θεώ. Μερικοί είπατε ότι είμαι πολύ φιλόδοξη. Είμαι. Εδώ πρέπει να επιλέξουμε σωστά τα πεδία μάχης. Ορισμένα από τα αξιότιμα μέλη αναφέρθηκαν στη βιοπικιλότητα. Και εγώ πιστεύω ότι η βιοπικιλότητα είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι η κληρονομιά μας. Είναι κρίσιμο για μας να διατηρήσουμε την κληρονομιά μας να εξασφαλίσουμε ώστε και οι παραδόσεις μας και οι αξίες μας και ο τρόπος ζωής μας να διατηρηθούν και η βιοπικιλότητα. Και όχι απλώς και μόνο επειδή υπογράψαμε, υπογράψαμε τις σχετικές συνθήκες για τη βιοπικιλότητα, αλλά γιατί είναι πραγματικά σημαντικό για όλες και όλους μας. Εξασφαλίζει ποιότητα ζωής. Από την ποικιλία και μες στις χώρες μας, αλλά και ανάμεσα στις χώρες μας. Αυτό το 7% του πρασινίσματος. Αυτό επίσης αποτελεί πρόβλημα για ορισμένους. Μία συζήτηση μπορεί να περιστραφεί γύρω από το ότι το 7% δεν θα πρέπει να είναι ανακμετάλλευση αλλά αναπεριφέρεια. Αυτό είναι μια δυνατότητα. Γιατί τότε παίρνει κανείς περιοχές, μεγαλύτερες περιοχές και να δημιουργηθεί βιοπικιλότητα εκεί στη βάση του 7%. Δεν λέω λοιπόν ότι ολόκληρη η Ιρλανδία θα πρέπει να καταλήξει την παραγωγή και να τα παράγουμε όλα στη Γερμανία. Θα πρέπει να είναι μικρότερες περιφέρειες, όχι χώρες ολόκληρες. Αλλά μια μικρή χώρα όπω η Δανία, εκεί όπου υπάρχει ας πούμε ένα ποτάμι. Εμείς έχουμε, δόξα τω πολλέ βροχές αυτέ τι μέρε. Έχουμε πρόβλημα βέβαια και λόγω της αλλαγής του κλίματος. Ωραία, εντάξει, ας φύγει λοιπόν η εκμετάλλευση, ας μπουν εκεί μερικές αγελάδες να βόσκουνε και να διασώσουμε κάπου την αρρώσιμη γη. Προτάσεις είναι αυτές. Ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να φωτίσουμε το θέμα και να το συζητήσουμε, να βρούμε δηλαδή διαφορετικούς τρόπους να ξεψαχνίσουμε την πρόταση της Κομισιόν και να δούμε πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Αυτά είναι θέματα προσυζήτηση που θα καταλήξουν δεν ξέρω. Μπορώ να σας υποσχεθώ βέβαια ότι θα κάνω κάθε τι το δυνατόν για να βρω κοινέ λύσεις για το μέλλον. Και θα διατηρήσω το διάλογο μαζί σας γιατί το είπα και στην αρχή και θα το ξαναπώ. Δεν έχουμε μόνο μια ιστορική ευκαιρία μπροστά μας, έχουμε και μια ιστορική ευθύνη να αναζητήσουμε κοινό έδαφος στην αγροτική μεταρρύθμιση. Και θέλουμε και πρέπει να το κάνουμε. Ας δουλέψουμε λοιπόν για να προχωρήσουμε την Ευρώπη μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μετ. Ήταν σαφέστατα όλα όσα μας είπε. Όλοι προβληματιστήκαμε, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την ειλικρίνειά σου, τη γνώση ε, σου γύρω από τα θέματα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Θα συνεργαστούμε με τη Δανέζικη Προεδρία για να βρούμε αυτό το κοινό υπόβαθρο, την κοινή πλατφόρμα. Ήταν μια πολύ καλή συζήτηση με διαφορετικές απόψεις φυσικά, αλλά και ένα κοινό πνεύμα που μας ενώνει σε αυτή τη μάχη. Λοιπόν, δύο λεπτά διακοπή για να χαιρετήσουμε την Προεδρεύουσα και θα συνεχίσουμε μετά άλλα δύο σημεία στην ημερήσια διάταξη. Pas, hein. Et comme on n'a pas d'hiver. Euh... C'est ça. Donc c'est en fait visiblement un moucheron qui. Colleghi, dobbiamo riprendere. Συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Σε facciamo veloce. Λοιπόν, αν κάνουμε γρήγορα, τελειώσουμε και πιο γρήγορα. Punto 11 Σημείο 11. Γεωγραφικές ενδείξεις των αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων. Χέρμπερτ Ντόρφμαν εισηγητής. Απλουστεύει την ισχύουσα ε, νομοθεσία με πέστερες ενδείξεις για την προέλευση και τις ετικέτες. Ο Χέρμπερτ Ντόρφμαν έχει το λόγο. Και αν θέλουν και οι εκπρόσωποι της Κομισιόν μπορούν να πάρουν το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσω Ιταλικά, ε, γιατί είναι καθαρά Ιταλικό το πρόβλημα μου φαίνεται. 70% των αρωματικών κρασιών στην Ιταλία παράγονται. θα έπρεπε όμως να εξηγήσω πώς έχει η κατάσταση. Είναι λίγο δύσκολη. Εμείς ως Επιτροπή πρέπει να κάνουμε μια γνωμοδότηση για όλο το κείμενο αλλά για ένα κομμάτι του κειμένου που αφορά στην ένδειξη προέλευσης δεν ε, γνωμοδοτούμε, αλλά είμαστε στην απόφαση ως Επιτροπή Γεωργίας. Θα ήθελα τώρα να, πω ότι τα αρωματικά κρασιά χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Το βερμούτ, με 16% αλκοόλ, αρωματικά κρασιά νορμάλ με 14,5% ενόπνευμα <clears throat> και μετά έχουμε τα απεριτίφ. όπου το 50% πρέπει να είναι αμπελινικά προϊόντα. Παραγωγή είναι κατά 70% η Ιταλία, μετά λίγο στην Ισπανία με τη Σαγκρία και μετά λίγο στη Γερμανία. Το Glühwein. Και δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα γύρω στην Ευρώπη. Με αυτή την περιγραφή. Τώρα, ε, πρόκειται για ευθυγράμμιση με τη Λισαβόνα. Η Κομισιόν προτείνει όλα τα ζητήματα αυτά ως ε, κατεξουσιοδότηση πράξης να δούμε τι θα κάνουμε σε αυτό. Τα αρωματικά κρασιά μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο με προσθήκη εινοπνεύματος... Ε, για να φτάσουμε στα ποσοστά. Βέβαια έχουμε και άλλες τεχνολογίες όπως είναι ε, κατάψυξη, απόσταξη ζαχάρωση. Πολυτεχνικά πράγματα. Σήμερα το βασικό κρασί πρέπει να είναι επιτραπέζιο κρασί, ευρωπαϊκό κρασί. Όταν λέμε απλώς κρασί, πρέπει να εννοούμε ότι πρόκειται για κρασί της Ευρωπαϊκής δεν λέμε ότι πρόκειται για κρασί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άμα λέμε απλώς κρασί μπορεί να είναι και εισαγόμενο κρασί από μη κοινοτικές χώρες. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κομμάτι που λέει ότι πρέπει να έχουμε γεωγραφική ένδειξη που την ξέρουμε από το κρεσί και για τα αρωματικά κρασιά. Αν πάρουμε εμείς το σύστημα παραγωγής ε, βλέπουμε ότι όλα αυτά τα αρωματικά κρασιά είναι στα χέρια της μεγάλης βιομηχανίας, π.χ. Μαρτίνι. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα ε, με τα αρωματικά κρασιά, με τα αρωματισμένα κρασιά, γιατί παράγονται με συνταγές πολύ ιδιάζουσες, τις οποίες γνωρίζει η βιομηχανία και οι οποίες δεν θα δημοσιοποιηθούν τις οποίες δεν θα δημοσιοποιούσε ποτέ για να τις ε, παράγουν άλλοι. Μπορεί να υπάρχει όμως ενδιαφέρον για τη σαγκρία ή ε, για διάφορα άλλα προϊόντα. Πρόκειται, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ε, για τη νέα νομοθεσία που μοιάζει με την νομοθεσία των κανονικών ε, Νομίζω ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ε, Κομισιόν. Η πολιτική συζήτηση θα πρέπει να ε, σταθεί κυρίως στην ευθυγράμμιση. Ευχαριστώ Ντόρφμαν. Έραντς Γκαρσία θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν για την ε, έκθεση που αφορά αυτή την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Προτείνει αναθεώρηση του συνόλου των κανονών για να διασαφινιστούν περισσότερο κάποιες έννοιες που αφοράν την ετικετοποίηση, τον ορισμό, την ε, προστασία των ε, περιοχών πάνω αυτά τα αρωματισμένα κρασιά, φαίνεται ότι αυτή η κατηγορία των ε, ε, αρωματισμένων αμπελονικών προϊόντων θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Στην χώρα μου τουλάχιστον η πρόταση αυτή έχει γίνει ευμενώς αποδεκτή, γιατί όπως είπατε η Ιταλία, η Γαλλία και η χώρα μου αφορώνται περισσότερο αυτήν την ιδέα. Η βελτίωση της ποιότητας και καλύτερη νομοθεσία για να βελτιωθεί η ποιότητα των ε, κρασιών που υποπέπτουν σε αυτή, υποπίπτουν συγγνώμη, σε αυτή την κατηγορία είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες επεξηγήσεις. Σε αυτό το νομοθετικό κείμενο θα πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να είναι σε θελούσια βάση η ιδέα της προσθήκης συνοπνεύματος. Είναι κάτι το οποίο ζητεί ή τη ζάχαρη φερρυπίνη για το βερμούτι. Είναι κάτι το οποίο το ζητά ο κλάδος και θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλείς κανόνες για να γίνονται τέτοιου ενέργειες. Ούτως ή άλλως σας θέλω να σας ευχαριστήσω για την θετική σας έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Ντόρφμαν που βρίσκεται στη φάση συντάξεως ε, της εκθέσεως. Έχω ορισμένες συμπληρωματικές ερωτήσεις. Διαβάζοντας το έγγραφο βλέπω ότι έχει πολλές ουσιαστικές λεπτομέρειες και αν κατανόησα καλά από τα όσα είπε ο κύριος Ντόρφμαν έχει να σχολιάσει ορισμένα από τα σημεία του εγγράφου του και άλλα όχι. Όμως στην εισαγωγική του έκθεση λέει ότι οι στόχοι και τα άλλα στοιχεία σχετικά με τους ορισμούς διατυπώσεις αλλά και επισημάνσεις των αρωματικών κρασιών καθώς και την προστασία των γεωγραφικών προελεύσεων αυτά θα πρέπει όλα να καθοριστούν από τον νομοθέτη. Το Κοινοβούλιο είναι νομοθέτης άρα πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε στην λήψη της αποφάσεως. Και βλέποντας παρακάτω στο άρθρο 14, βλέπω για παράδειγμα ένα θέμα τώρα το οποίο επέλεξα και που αναφέρεται σε εθνικές διαδικασίες και όπου λέει είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης να απορριφθεί μια γεωγραφική προέλευση εφόσον δεν εκπληρώνται ορισμένε προϋποθέσεις. Αυτό πάντως το έγγραφο για μένα ανοίγει πολλά ερωτηματικά και διορωτώ πού εντοπίζονται τα νέα στοιχεία. Για παράδειγμα για τις ε, ονομασίες γεωγραφικής προελεύσεως, ε, αυτό προκύπτει από τον κανονισμό για τα κρασιά. Στη διαδικασία αυτή πού μπορούμε να τροποποιήσουμε κάποια πράγματα. Είναι απλώς τεχνικού χαρακτήρα που ε, θα πρέπει βέβαια να μιλήσει μονάχα για τα κατεξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις. Και αν στον τομέα αυτό υπάρξουν τροποποιήσεις, για παράδειγμα στο άρθρο 14 θέλω να ρωτήσω ποιος καθορίζει τις ιδιαίτερες αυτές απαιτήσεις και τι περιλαμβάνουν αυτές οι απαιτήσεις. Αυτά είναι καθορισμένα ήδη στον κανονισμό αγοράς του κρασιού ή ανοίγουμε εδώ ένα νέο πεδίο και εφόσον ανοίγουμε νέο πεδίο τότε νομίζω το Κοινοβούλιο έχει το καθήκον να εγγύψει τις λεπτομέρειες και να συναποφασίσει. Άρα πρώτα να τη συζητήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρόταση της Επιτροπής για αναθεώρηση είναι σε θετική κατεύθυνση. Θέλω να σημειώσω ως ε, ιδιαίτερη σημασία ε, την ε, πρόθεση στη χρήση του ίνου προς βελτίωση της ποιότητας των αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων ε, πράγμα που μας ενδιαφέρει απόλυτα γιατί δημιουργεί άλλη μία ε, διέξοδο για τη διάθεση του προϊόντος. Βεβαίως ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε τις συνθήκες διάθεσης του ευρωπαϊκού ίνου. Νομίζω ότι είναι επίσης θετικό να αναφερθούμε στην αναγνώριση της τεχνολογικής εξέλιξης της τελευταίας 20 που επιτρέπει την εγγύηση της ποιότητας αλλά και τη διαφεροποίηση του προϊόντος ε, παράλληλα με τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, ε, είναι ε, χρήσιμο να αναφέρουμε ότι όσον αφορά τον καταναλωτή, η διασφάλιση της ακριβούς ενημέρωσης και ποιότητας που δίνει και ιδιαίτερη σημασία στον παραδοσιακό χαρακτήρα του τρόπου παραγωγής αλλά και της παρουσίας αυτών των προϊόντων είναι κάτι το οποίο βελτιώνει τη σχέση του προϊόντος με τον καταναλωτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο Δόκτωρ Τζορίλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω μετά από αυτά που είπε ο Έλληνας Ευρωπαϊκός βουλευτής ότι ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ενημερώσουμε την πολύ παλιά νομοθεσία που υπάρχει ώστε να είμαστε σίγουροι ότι περισσότερα είδη κρασιού μπορούν να προσθεθούν σε αυτά τα προϊόντα και ότι οι ορισμοί ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις απαιτήσει της αγοράς. Ώστε, ενώ σήμερα έχουμε προϊόντα με χαμηλό βαθμό ε, που συμπεριλαμβάνονται εδώ και μετά από συζητήσεις που έχουμε με τη βιομηχανία και τους ενδιαφερόμενους να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές προς τις απαιτήσει της αγοράς ώστε περισσότερα είδη κρασιών αν θέλετε να μπορούν να υποπίπτουν σε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Α, όχι, κι άλλος θέλει το λόγο. Χέρμπερτ. Επανέρχομαι, λέει η κυρία Κλάς, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναπαραπομπή αυτής της οδηγίας στο Κοινοβούλιο τίθεται υπό συζήτηση. Εάν υπάρχει συνολική αναδιατύπωση του κανονισμού, τότε υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο συζητήσεως. Τα αρωμα, αρωματισμένα ποτά, τα οποία γεμίζουν τα μπουκάλια σε διαφορετικές περιφέρειες και εκεί πρέπει να είναι σωστή και η επισήμανση και πρέπει βέβαια να προσέξουμε και πάρα πολύ τις επισημάνσεις γεωγραφικής προελεύσεως. Και τι θα πει εμφιαλωμένο στο τάδε μέρος. Αυτό το εμφιαλωμένο πρέπει να μπαίνει με μεγάλα στοιχεία για να φαίνεται καθαρά. Λοιπόν, ε, ο, ο τρόπος με τον οποίο θα χειριστούμε το έγγραφο, αυτό θέλω να μάθω. Ε, μπορούμε να κάνουμε ε, τροποποίησεις, ναι ή όχι. Δόκτωρα Τζορίλα, θέλετε να μιλήσετε, μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντόρφμαν για να τελειώνει. Σε αυτό το σχέδιο πρόταση υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο είναι καινούριο σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό που είναι το τμήμα που αφορά την γεωγραφική προέλευση. Διότι παλιά υπήρχαν μόνο τέσσερα ονόματα, τώρα ευθυγραμμίσαμε αυτό το κανονισμό με σε, τους άλλους κανονισμούς που αφορούσαν υνοπνευματόδη προϊόντα και κρασιά και τις περιφέρειες στις οποίες παράγονται στην Ευρώπη. Αυτό το κάναμε ώστε όσον αφορά την γεωγραφική ένδειξη για τα αρωματοποιημένα αμπελονικά προϊόντα να τα ευθυγραμμίσουμε όπως σας είπα με τους άλλους κανονισμούς και να τα εναρμονίσουμε. Τώρα, εάν με ρωτάτε, εάν μπορεί κανείς να παρέμβει, το Κοινοβούλιο μπορεί να παρέμβει. Φέσαμε το θέμα στο Συμβούλιο και σε εσά και όπως σας είπα, Πρόκειται για επικαιροποίηση παλαιού κανονισμού με τις γεωγραφικές ενδύσεις. Υπάρχουν πολλέ αλλαγέ όσον αφορά τον ορισμό, αλλά βεβαίω έχει το δικαίωμα να προτείνετε αλλαγέ. Και έχουμε εδώ και κάποιον από την νομική υπηρεσία της Γενικής μου διεύθυνση. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μου ε, το επιβεβαιώνει, βεβαίως και μπορείτε να υποβάλλετε αλλαγές. Ευχαριστώ. Χέρμπερτ, τα συμπεράσματα. Ίσως προηγουμένως να μην διατύπωσα τις σκέψεις μου με ιδιαίτερη ακρίβεια, γι' αυτό επανέρχομαι στο ερώτημα της κυρίας Κλάς. Το περιεχόμενο του εγγράφου όντως χωρίζεται σε δύο τμήματα σε ό,τι αφορά τη δική μας αποφασιστική αρμοδιότητα. Το πρώτο μέρος, όπου αναφέρεται στην παραγωγή των προϊόντων αυτών, αυτό είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και εκεί ο εισηγητής είναι ο κύριος Μπαρτολότσι που είναι τρεις σειρές πίσω μου και είναι και νέος συνάδελφος εδώ και θα συντάξει γνωμοδότηση. Για το δεύτερο μέρος, για τις γεωγραφικές ενδείξεις, είμαστε αρμόδιοι επί της εμείς, η δική μας Επιτροπή. Βεβαίως σε διαδικασία συναποφάσεως, άρα ασφαλώς και έχουμε συναποφασιστική αρμοδιότητα εμείς στο Κοινοβούλιο δηλαδή. Για τη δεύτερη ερώτηση της κυρίας Κλάς, τα νέα στοιχεία δηλαδή, νομίζω απήντησε ο ίδιο ο κύριος Σορίλα και δεν ε, έχω τίποτε παραπάνω να πω. Ήθελα πάντως να παρακαλέσω όλες και όλους τους συναδέλφους, όσοι ενδιαφέρονται δηλαδή για το θέμα, να έρθουν σε επαφή μαζί μου, ώστε τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να συντάξουμε μαζί μια ε, καλή γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου μας. Ευχαριστώ τον Χέρμπερτ Ντόρφμαν. Πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καλό λοιπόν εδώ στο Προεδρείο τον ανεξάρτητο Πρόεδρο του Συμβουλίου της ΦΑΟ, τον ε, κύριο ε, Λουκ Γκιό, που θα μας μιλήσει για την ε, τροφιμική ασφάλεια. Κύριε Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκαν πολλές φορές για την τροφιμική ασφάλεια και Ιταλικά μιλάτε, έτσι δεν είναι. Έλεγα λοιπόν κύριε Πρόεδρε ότι η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκαν πολλές φορές για το θέμα της τροφιμικής ασφάλειας και ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Ξέρουμε ε, ότι ε, η αύξηση των εισοδημάτων σε πολλές ε, περιοχές του κόσμου και αύξηση του πληθυσμού από τα 7 στα 9 δις μέχρι το 2050 χρειάζονται αύξηση της παραγωγής. Η έκθεσή μας ε, που ψηφίσαμε εδώ του κυρίου Σάρμπο στην Επιτροπή μας για το 2010 υπογραμμίσαμε την ανάγκη για να διασφαλίσουμε την τροφιμική ασφάλεια στην Ευρώπη προσφέροντας στους καταναλωτές σίγουρα τρόφιμα ψηλής ποιότητας με λογικές τιμές και εγγυόμενοι το γεωργικό εισόδημα. Πρόκειται για τους κεντρικούς στόχους της ΚΑΠ που όπως γνωρίζετε τώρα είναι και το βασικό θέμα συζήτησης αυτό το δεύτερο τμήμα της Γεωργίας. Είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν όλους μας και πρέπει να ακολουθήσουμε τη γνώμη σας και την έκθεσή σας. Σας δίνω λοιπόν ευθύς αμέσως το λόγο κύριε Πρόεδρε Γκριό και ελπίζω να έχουμε και ενδιαφέρουσα συζήτηση μετά την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, διότι μου δίνετε τη δυνατότητα να λάβω το λόγο σήμερα στην Επιτροπή σας και να σας μιλήσω για ένα τόσο σημαντικό θέμα, όπως αναφέρατε, την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση στα πλαίσια της ε, ασφάλειας των ειδών διατροφής. Η Επιτροπή σας, στην οποία θα πρέπει να προσθεθεί και η Αλία, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, αυτού του θέματος. Εμένα με εξέλεξαν μυστική πληροφορία, ε, συγγνώμη, ψηφοφορία, τα 191 κράτη-μέλη της οργάνωσης τον Νοέμβριο του 2009 και για διάρκεια της πρώτης θητείας μου επισκέφθηκα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο τον προηγούμενο χρόνο. Συνάντησα κάποιους από εσά και έκανα τις πρώτες ανταλλαγές απόψεων για το σχέση μεταξύ ΦΑΟ και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 12 μήνες μετά από αυτή την πρώτη συνάντηση υπάρχουν τόσο μεγάλες εκτενές που, εξελίξεις που μου φαίνεται ότι είναι εντελώς απαραίτητη και σκόπιμη να έχουμε μία νέα συνάντηση για να σας ενημερώσω για δύο λόγους για τις αλλαγές. Πρώτα απ' όλα, διότι πρέπει να σας πω ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην έδρα της ΦΑΟ στη Ρώμη και δεύτερον, για να μου πείτε εσείς ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Με την επανεμφάνιση του λιμού και της ένδυας σε μεγάλη κλίμακα στο περιοχή του κέρατος της Αφρικής το 2011 δυστυχώς επιβεβαίωσε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η ασφάλεια των ειδών διατροφής θα είναι για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ένα από τα ουσιώδη θέματα με τα οποία θα πρέπει να ασχολείται όλος ο κόσμος. Τα μέλη του G20 το κατάλαβαν και μπόρεσαν να εγκρίνουν ένα ειδικό σχέδιο δράσης. Θα πρέπει να σας πω ότι το 1950 είμαστε 2,5 δις άνθρωποι στον κόσμο και το 2050 προβλέπεται ότι θα είμαστε 9. Στο χρονικό λοιπόν αυτό διάστημα μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε η διατροφή για τέσσερα δις περισσότερο Δεν ξέρω όμως αν θα συνεχίσει κάποιο τέτοιο να γίνει. Αυτό που σας είπα το κατάλαβαν τα μέλη του G20 και για τη διάσκεψη αρχών κρατών και κυβερνήσεων για τον, τον Νοέμβριο ενέκριναν ένα ειδικό σχέδιο δράσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα της Επιτροπής σας πρέπει να πω ότι συμμετείχε σε όλη αυτή τη διαδικασία του σύναγγης. Εάν λάβω υπόψη τις συζητήσεις που έγιναν στην Ολομέλεια και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο που αφορά την αλυσίδα διανομής των ε, γεωργικών προϊόντων, τα διοκτώνα και την ε, κατασπατάληση των ειδών διατροφής ή αν λάβω υπόψη τις παρεμβάσεις που έγινε συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ε, ε, βοήθειας και συνδρομής των πλέον ενδεών που έγινε εδώ και μερικές εβδομάδες. Στη Ρώμη, η πιο πρόσφατη και βεβαίως αυτή που θα έχει περισσότερες ε, επιπτώσεις, εξέλιξη για την ζωή και αποδοτικότητα της οργάνωσής μας για την καταπολέμηση της πείνας είναι ότι έχουμε ένα νέο γενικό διευθυντή, τον κύριο Ζωζέ Γκρατσιάνο Ντασίλβα από την Βραζιλία, από την 1η Ιανουαρίου. Και πρέπει να πω ότι οι προηγούμενοι γενικοί διευθυντέ έμειναν για πάρα πολύ καιρό στην οργάνωσή μα. Οι πρώτε του δηλώσει του γενικού μα διευθυντή αποδεικνύουν ότι πραγματικά θέλει να υπάρξει μία αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας στο ΦΑΟ που τη χρειάζεται πάρα πολύ ώστε να υπάρξει εκ νέου αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και εντός και εκτός της οργάνωσης και να γίνουν ε, οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή όλα τα σχέδια μεταρρύθμισης που εγκρίθηκαν το 2008. Όλοι ξέρουμε ότι και οι καλύτερες μεταρρυθμίσεις δεν, ε, ε, εάν δεν εφαρμόζονται σωστά, δεν είναι επιτυχής. Ο ε, νέος λοιπόν Γενικός Διευθυντής σίγουρα θα προσθέσει με τον δυναμισμό του όσον αφορά την αλλαγή αυτών των διαδικασιών που σας ανέφερα. Η μεταρρύθμιση της Επιτροπής για την Παγκόσμια ασφάλεια των ειδών διατροφής που ε, απευθύνεται και στην ε, κοινωνία των πολιτών και στο Συμβούλιο βασίζεται σε αυτή την διαδικασία της αποκέντρωσης έχει σχέση με τις διάφορες περιφερειακές διασκέψεις και αποτελεί ένα από τα πλέον ορατά στοιχεία της αλλαγής των διαδικασιών που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτής της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Το 2012 ο νέος Γενικός Διευθυντής θα ολοκληρώσει αυτό το στάδιο και θα περάσει στο επόμενο. Η, στα πλαίσια αυτά η συνεργασία νότου-νότου είναι ένας από τους πέντε άξονες στρατηγικής για την ΦΑΟ. Και βεβαίως αυτό δεν ε, αποκλείει ότι θα υπάρξουν ε, και άλλες ε, δράσεις συνεργασίας μεταξύ Νότου και Βορρά. Όσον αφορά την πιο μεγάλο άνοιγμα προς την κοινωνία των πολιτών και την συμπερίληψη του ιδιωτικού τομέα, πρέπει να πω ότι εφέτος θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα των συνεταιριστικών. Στον τομέα της επικοινωνίας προς τα έξω και προς τα μέσα έχουν γίνει πάρα πολύ μεγα... ετοιμάζονται πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην ΦΑΟ και τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Άλλα σημαντικά θέματα όπως ε, η θέσπιση ε, νέων ε, ε, θελούσιου χαρακτήρα οδηγιών για το δικαίωμα στην σύντηση, οι γενικές γραμμές που αφορούν τα, τα καθεστώτα εγγύου ιδιοκτησίας βρίσκονται σε τελικό στάδιο στη Ρώμη καλύτερη συνεργασία μεταξύ όλων των οργανώσεων των Ηνωμένων Εθνών είναι κάτι το οποίο αναμένουμε επίσης. Άρχισαν τέτοιου είδους κινήσεις, αλλά θα πρέπει να ενταθούν και η δημιουργία συνεργειών πιο ισχυρών είναι απαραίτητη όρη και προϋποθέσεις για να επιτύχουμε. Απαραίτητα, ε, αναμφίβολα, συγγνώμη, κ. Γκρατσιάνο σύντομα θα επισκεφθεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εταίρος της ΦΑΟ. 42% του προπολογισμού έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Θα σας ανακοινώσει το μήνυμά του και σήμερα εγώ δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες που θα πει, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες σκέψεις άτυπα. Η θέση μου, όπως ξέρετε, είναι στο κέντρο των συζητήσεων που γίνονται μεταξύ κρατών μελών, γραμματείας της οργάνωσης και σύνολο των ε, συνομιλητών και εταίρων. Όπως είπα και πέρσι στο Στρασβούργο, θα μπορούσε η ανάπτυξη των σχέσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να βασιστεί σε δύο άξονες. Πρώτα απ' όλα, κοινέ σκέψεις για θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της προβληματικής για την ασφάλεια των ειδών διατροφή. Το να μοιραστούμε εμπειρίες και να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων και αναλύσεων και δυνατών λύσεων δεν μπορεί παρά να μας βοηθήσει στο να επιλύσουμε το πρόβλημα που μας απασχολεί που είναι η καταπολέμηση της πείνας. Για να αναφέρω ένα παράδειγμα, στα πλαίσια της ΚΑΠ και της ε, εξέλιξής της, είναι σαφές ότι οι περισσότερες βασικές αρχές θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σήμερα στα πλαίσια του, των περιφερειακών γεωργικών πολιτικών για όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Όσον αφορά την, ΚΑΠ του 2013, οι επιπτώσεις της για την ε, παγκόσμια ασφάλεια των ειδών διατροφής και τις παγκόσμιες αγορές θα μπορούσε να εξηγηθεί καλύτερα και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει σε όλους να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεύτερος άξονας, καλύτερη ε, εξήγηση και έκφραση του τι ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα όργανα διακυβέρνησης της ΦΑΟ. Δεν ε, αγνοώ την κατανομή των ρόλων και των ε, ε, εντολών που υπάρχουν μεταξύ ε, Συμβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εξωτερικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των κρατών μελών. Ξέρω ότι υπάρχουν περιορισμοί, αλλά θα πρέπει να τους ξεπεράσουμε ώστε να μπορέσει να μιλήσει με ενιαία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διεθνές επίπεδο και το ε, γεωργικό κοινοβούλιο του πλανήτη, όπως λέγει και ο Επίτροπος Μπαρνιέ που αποτελεί η ΦΑΟ και τα διάφορα όργανα της. Σήμερα στη ΦΑΟ δεν υπάρχει σε πολιτικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε επίπεδο συνεισφοράς της. Χρειάζεται ε, η παρουσία της να γίνει πιο ορατή και πιο ενεργή σε υψηλό επίπεδο, διότι όπως απεδείχθη και στο παρελθόν, στην ε, ΦΑΟ μπορείτε εσείς να διασφαλίσετε το διάλογο με διάφορες περιφερειακές ομάδες. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο. Είναι ένα ζήτημα αυτό το θέμα της τροφιμικής ασφάλειας. Πρέπει να ε, ε αναρωτηθούμε ε, και να προβληματιστούμε πολύ σοβαρά γύρω από όλα αυτά λόγω των στενών δεσμών που έχει όλη αυτή η ιστορία και με την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ο κύριος Σεγκοβιέσκη, ο, πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος. Μάλλον ο κύριος Γκαρόν πρώτα. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία υπόθηκαν και πιο συγκεκριμένα στην ιδέα ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε, να στείλουμε ένα διπλό μήνυμα. Και αυτό λόγω της ανησυχίας που έχουμε για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον με την τροφιμική ασφάλεια. Αλλά και τρέφοντας επίσης ε, την ε, ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε μια κατάσταση αυτού του τύπου. Γι' αυτόν τον λόγο την προηγούμενη εβδομάδα εμείς εγκρίναμε ε, στο Κοινοβούλιο μια έκθεση για την σπατάλη, για την σπατάλη στα τρόφιμα. Εγώ θα ήθελα να ξέρω εάν υπάρχει πρωτοβουλία εκ μέρους ε, της ΦΑΟ, εάν, τι προτεραιότητες ε, έχει σχετικά αυτό το θέμα, διότι έχω την εντύπωση ότι αυτό το θέμα κάπου το είδαμε περιθωριακά. Ένα θέμα το οποίο το αναθέσαμε σε μερικές φιλανθρωπικές οργανώσεις και όχι ως κάτι το οποίο αμφισβητεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο ε, παρα, ε, δημιουργεί αρνητικά ε, μοντέλα. Διότι εδώ πρόκειται για σπατάλη ε, τροφίμων απολύτως ε, βροσίμων. Ο Βοράς, το πλούσιο κομμάτι του κόσμου στην Ευρώπη, αρκετά εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και υποφέρουν από και το ίδιο αντιμετωπίζει και η Νότια Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και από το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τη ΦΑΟ. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει βούληση για συνεργασία σχετικά. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρόνα για αυτή την τοποθέτηση. ενημερώθηκε και ο πρόεδρος ε, της ΦΑΟ για την έκθεσή μας σχετικά με την έκθεση που έχουμε εγκρίνει. Ο πρόεδρος Εκερέσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. γίνεται μεγάλη προσπάθεια να δημιουργηθούν οι ρυθμίσεις οι οποίες θα έχουν παγκόσμια ισχύ. Έχουμε στην Ευρώπη την προσπάθεια ρύθμισης χρηματιστηριών και τραπεζών και γίνεται μια προσπάθεια παγκόσμιας δραστηριοποίηση. Έχουμε και τον ΦΑΟ με ιδιαίτερη εξειδίκευση και ο οργανισμός αυτός σε όλη την ιστορία έπαιξε σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση της στόχιας και της κακής σύντησης. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση και ρωτώ ποια κατά τη γνώμη σας θα είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την γεωργική παραγωγή. και διαρθρωτικά και γεωγραφικά. Δηλαδή, τι παραγωγή θα έχουμε, τι τρόφιμα θα παράγονται, θα αλλάξει το καταναλωτικό μας πρότυπο. και θα μειωθεί η δράση του κερδοσκοπικού κεφαλαίου στην αγορά τροφίμων. Γιατί πρόσφατα η κρίση στα τρόφιμα δεν έγινε ίσως τόσο αισθητή στην Ευρώπη, έγινε όμως έντονα αισθητή παγκοσμίω, ως αποτέλεσμα όχι μόνο αντικειμενικών συνθήκων, αλλά και λόγω κερδοσκοπίας. Η παρούσα κρίση, παγκόσμιο χαρακτήρα που αντιμετωπίζουμε τώρα, πώς άπτεται της ασφάλειας τροφίμων. Και ποιες δράσεις αναλαμβάνονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν άλλη προσέγγιση, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία διαφορετική προσέγγιση και τέλος άλλη πάλι είναι η προσέγγιση στην Ευρώπη. Θέτω βέβαια πολλές ερωτήσεις, αλλά ίσως είναι περισσότερο σχόλια παρά ερωτήσεις. Και βέβαια η απελευθέρωση του εμπορίου, από την οποία όλοι κερδίζουμε, διότι εξασφαλίζει μεγαλύτερη ασφάλεια τροφίμων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και προβλήματα με τις προδιαγραφές, πρότυπα. Δηλαδή πάντοτε πρόκειται για μια ανταλλαγή. Δηλαδή, πάντα δίνει κανείς κάτι για να αποκτήσει κάτι. ή να δουν και λαβίνα. Αυτό θα μπορούσε να καταστεί σαφέ και με ένα πίνακα. Πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρος Μπολε, ε, Μποβέ, συγγνώμη στο λόγο. Θα πω Λουκ, δεν θα πω μισιο γιατί αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, όλοι οι Γάλλοι μας γνωρίζουν, ε, το, το ξέρουν, οπότε μπορούμε να, μιλάμε, να, να μην μιλάμε με το ΣΥΣ και με το σας, αλλά με το εσύ. Λοιπόν, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση αρκετά πολύπλοκη σε διεθνές επίπεδο, το εξήγησες γενικώ, θα ήθελα να θέσω τρία σημεία. Οι, ε, οι συζητήσεις δηλαδή αποτυχία δεν κατέληξαν μεταξύ των άλλων δηλαδή η αιτία της αποτυχίας είναι και η Γεωργία. Δεν θα ήταν πλέον καιρός σήμερα να βρούμε ένα άλλο μέσο εμπορίου για τη γεωργία σε διεθνές επίπεδο από ότι αυτή η αρχαϊκή μέθοδος που έχει επιβληθεί στην ΠΟΕ πρέπει να βγούμε έξω από αυτή τη, τη λογική. Πόσο μάλλον δηλαδή που Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερο να διαπραγματευτούμε μέσα από πολυμερείς συμφωνίες και όχι μέσα από αυτές τις διμερείς συμφωνίες. Βλέπετε τι γίνεται με το Μερκοσούρ, τα προβλήματα που θα τεθούν και η γεωργία θα, θα χρησιμοποιηθεί ως αντάλλαγμα για, για, για τις υποχωρήσεις υπηρεσίες και στη βιομηχανία. Το ίδιο θα συμβεί και με το Μαρόκο. Δηλαδή ξέρω ότι η ΦΑΟ κάνει συγκεκριμένες έρευνες για το πού προρίζονται ε, οι διάφορες εκτάσεις ε, και το land graving όπως λένε στα αγγλικά. Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή σε πολλές περιοχές του κόσμου. Έχω κατά νου την Αφρική και όχι μόνο την Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα μεταξύ των κρατικών πολιτικών ή των επιχειρησιακών πολιτικών και με απόγειο την ιστορία των αγροκαυσίμων που υποσκάπτουν όλη τη λογική της τρόφιμικής γεωργικής παραγωγής. Τώρα για το θέμα των σχέσεων νότου-νότου και της ε, τριγωνικής σχέσης, πώς προχωράει αυτή η ιδέα να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υπηρετικούς ή πόλους που θα μπορούσαν να αποτελέσουν και το μόνο τρόπο για να προχωρήσουμε. Θα μπορούσες να μας πεις κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Ο Μάρτιν Χόσλινγκ. Ναι. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο μου ο Ζωζέ Μποβέ και νομίζω ότι η δυναμική των αγορών θα εξαρτηθεί στο μέλλον από την πορεία των καυσίμων, των βιολογικών καυσίμων που πάει να πει ότι θα χρειαζόμαστε περίπου 30 εκατομμύρια εκτάρια μόνο για την παραγωγή βιολογικών καυσίμων και πέρα από το βιοαέριο. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερα τολμηρό να πει κανείς ότι μπορούμε να ταΐσουμε σήμερα 7 δισεκατομμύρια ψυχές και σε 30 χρόνια θα μπορούμε να ταΐσουμε 9 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αν συνεχίσουμε έτσι με τη χρήση της γης αποκλείται να τα καταφέρουμε. Πρέπει στη διεθνή συζήτηση αυτά τα πράγματα να μπουν πολύ περισσότερο στο προσκήνιο. Αν δηλαδή ταιριάζουν, συντεριάζουν αυτοί οι στόχοι. Οι περισσότερες ε, γέε που πέφτουν θύμα του land grabbing, της αρπαγής των γεών δηλαδή σήμερα, ε, εξυπηρετούν και την παραγωγή καυσίμων ή διπλή χρήση όπως της σόγιας. Αυτό να μην το λησμονούμε. Και είπαμε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική έχει σημαντικές επιπτώσεις και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μελλοντική προμήθεια τροφίμων. Αλλά τι είδους ευρωπαϊκή πολιτική θέλετε, αν μπορούσατε να μας συμβουλεύσετε ανεξάρτητα, τι θα μπορούσατε να μας συμβουλεύσετε, δηλαδή προς τα πού να κινηθούμε. Γιατί εμείς λέμε ότι θέλουμε φιλοπεριβαλλοντική γεωργία, κάτι το οποίο εγώ υποστηρίζω σε πολλές, από πολλές πτυχές. Τώρα, τι ρόλο παίζει η Παγκόσμια Έκθεση Γεωργίας ως βάση για την περαιτέρω, παραπέρα δράση σας ή βασίζεστε περισσότερο σε μια γεωργία που θα χρειάζεται περισσότερες εισρωές στις βιομηχανικές χώρες για να παραγάγει και περισσότερο. Εμάς, ε, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει περισσότερο να ενισχυθούν οι μικροί παραγωγή στις φτωχές χώρες για να λυθεί το πρόβλημα της ε, προμήθειας τροφίμων επιτόπου και να απαλληλθούν έτσι οι επιπτώσεις των ε, ε, προβλημάτων που έχουμε προκαλέσει εμείς με την εντατικοποίηση της γεωργίας. Και είναι γνωστό ότι οι μικροί γεωργοί δεν μπορούν να αντέξουν στην παγκόσμια ανταγωνιστική γεωργία. Αυτό κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη λαμβάνετε, το λαμβάνετε εσείς υπόψη δηλαδή στην ε, διαμόρφωση πολιτικής σας. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες και μετά κύριο Σάγνιο. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον τα σχόλιά σας για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς δεν παίζει ρόλο στην πραγματικότητα μέσα στον ΦΑΟ και πώς θα μπορούσε να παίξει μεγαλύτερο ρόλο. Για πέστε λίγα περισσότερα γι' αυτό πώς βλέπετε να μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή και ποιες επιπτώσεις και συνέπειες θα έχει η αυτή η μεγαλύτερη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ κοίταξα και την ιστοσελίδα σας του ΦΑΟ δηλαδή και πολλά από τα θέματα που βλέπω να σας απασχολούν μας απασχολούν και μας εδώ δηλαδή η αλλαγή του κλίματος, ο ρόλος των συνεταιρισμών και άλλων οργανώσεων παραγωγών. Εσείς τον ΦΑΟ μιλείτε για τη σημασία που έχουν αυτά για τον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά αυτά περιλαμβάνονται και στη δική μα μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Βλέπω λοιπόν να υπάρχει επικάλυψη συμφερόντων μεταξύ των γεωργών μα, είτε είναι του αναπτυσσόμενου είτε είναι του αναπτυγμένου κόσμου. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι το εξή. Για χρόνια λέω εγώ και με υποστηρίζουν και άλλοι συναδελφοί μου και εδώ αλλά και στην Ολομέλεια ότι η αγροτική ανάπτυξη είναι κρίσιμη για τις χώρες εκείνες που έχουν ελλείψεις τροφίμων και που στην ύπεθρό του έχουν μέχρι και 95% του κόσμου που έχουν πρόβλημα να εξεύρουν τρόφιμα, να φάνε. Χαίρομαι που η Κομισιόν έχει αλλάξει τον προσανατολισμό της ε, αναπτυξιακής βοήθειας και προσφέρει περισσότερη ενίσχυση στη γεωργία. Γιατί εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την πολιτική μας εμπλοκή με τον ΦΑΟ αλλά και να μας πείτε επίσης ποιες επιπτώσεις θα έχει η μη συμμετοχή της Ευρώπης. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι εδώ χρειάζεται ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να δοθεί προς πάσα κατεύθυνση. Και βεβαίως σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Thank you, uh, Δεν πιστεύω να είμαι ο μόνος που θεωρώ ηρωνία στις τελευταίες δύο συζητήσεις που γίνονται σήμερα το απόγευμα εδώ, διότι μόλις πριν από μια ώρα μιλούσαμε για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φύγει ε, αγροτική γη από την παραγωγή τροφίμων. Και τώρα μιλούμε βέβαια για την ασφάλεια των τροφίμων και πολλοί είναι οι άνθρωποι στην Ένωση που μιλάνε, που πεινάνε, συγγνώμη. Ίσως να μην κατάλαβα καλά από τη μετάφραση, αλλά μου φάνηκε ότι είπατε τα τελευταία 20 λεπτά ότι 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουν από υποσυτισμό. Μήπω ήταν 8 εκατομμύρια, βέβαια μόνο οι διερμηνείς το γνωρίζουν αν ήταν 88. Αν είναι πράγματι 80 εκατομμύρια και αν είναι πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ παράξενος ο ορισμός του υποσυτισμού. Μήπως είναι παραπάνω από 25 μίλια από ένα McDonald's, διότι αυτό μου φαίνεται πραγματικά πάρα πολύ παράξενο και γελίο. Ο Χόισλινγκ πριν μίλησε για τα βιολογικά καύσιμα. Δεν συμφωνώ συχνά μαζί σου, Μάρτιν Χόισλινγκ. Μάλιστα, αν συμφωνήσω, θα αρχίσω να ανησυχώ και θα πω στον γιατρό. Αλλά βρίσκω ότι είναι σωστό αυτό που είπε. και η μεγάλη ε, δυσκολία εδώ είναι αν επανέρχεται στο, στα 1980 όπου ε, εκτοξευόταν η παραγωγή τροφίμων με σιτηρά τα οποία σάπιαν αποθήκες και είχαν πει ότι με τα πλεονάσματα αυτά που έχουμε του σταριού κάτι άλλο πρέπει να τα κάνουμε. Βρέθηκε μετά η τεχνολογία για να γίνουν αυτά τα πράγματα ενέργεια. Αυτά βέβαια χρειάστηκε χρόνο για να δημιουργηθούν τα σχετικά εργοστάσια κλπ. Φτάνουμε λοιπόν τώρα σε μια κατάσταση όπου έχουμε τα εργοστάσια αυτά και αυτά τώρα ζητάνε πρώτη ύλη. Είναι πολύ δύσκολο να πούμε ωστόσο ποια θα είναι η σοδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη, πόσε θα είναι οι σοδιές. Αν όμω υπάρχουν πλεονάσματα, πρέπει κάπου να διοχετεύονται για να μην πέσουν οι τιμές τόσο πολύ για τους αγρότες που να απογοητευτούν, να αποθαρρυνθούν και να σταματήσουν να παράγουν. Η λύση δεν είναι να αρχίζουν και να πάθουν να λειτουργούν τα εργοστάσια αυτά. Ωστόσο, Μάρτιν, νομίζω καλά έκανε και το είπε και είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει. Ωραία. Ο Μισελ Νταντά και μετά παρακαλώ να ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Λυκειό. Πέρυσι είχαμε μία διεθνή συνειδητοποίηση του θέματος της διαχείρισης των αποθεμάτων και της διαφάνειας αυτής της διαχείρισης και αυτό ως απάντηση στην παγκόσμια διακύμανση των ε, τιμών. Ε, η ΦΑΟ ε, συμμετείχε σε αυτήν την διαδικασία. Διαπιστώνει σήμερα μετά από τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ένα σχετικό άνοιγμα ή τίποτα δεν άλλαξε. Οπότε η διαχείριση των αποθεμάτων παραμένει ένα θέμα εθνικής στρατηγικής της κάθε χώρας και οι ελπίδες που δείξαμε για τις διάφορες λύσεις ε, δίνουν ελπίδα ή πρέπει να εργαστούμε προς άλλη κατεύθυνση. Ευχαριστώ Μισελ. Η δόκτωρ Μίτσι έχει το λόγο. Um, from Ο Δόκτωρ Μίτσι λείπει σε άλλη συνεδρίαση και έτσι εμένα. Ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Για την ώρα απλώς θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Άγνιου για την παρουσία του εδώ και τον κύριο ε, μάλλον για την παρουσία του εδώ και παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτησή σας. Ευχαριστώ την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Νομίζω ότι είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σου δίνω και πάλι το λόγο αγαπητέ Γκουγιό, λέει ο πρόεδρος, και θα ακούσουμε τις τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που κάνατε. Πριν απαντήσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξής. Η είναι μια οργάνωση που ανοίξει το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών που δεν έχει την δυνατότητα να υποχρεώσει τα κράτη να κάνουν κάτι και δεν μπορεί να θεσπίσει καμία πολιτική αν δεν συμφωνήσουν και τα κράτη-μέλη. Βεβαίω όλα αυτά γίνονται αν υπάρξει συνένεση. Συμφωνία μεταξύ όλων. Ξέρω ότι και εδώ οι συζητήσει δεν είναι πάντα εύκολε, αλλά κάποια στιγμή ο πρόεδρο χτυπάει το κουδουνάκι, εκεί βλέπουμε ποια είναι η πλειοψηφία. Σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι προσπάθεια μπορούμε ώστε να καταλήξουμε τελικά σε συνένεση. Συνένεση η οποία επιτυγχάνεται τελικά μέσα τη συμφωνία όλων, εκτός από κάποιους που δεν συμφωνούν αλλά σιωπούν. Έτσι λοιπόν παίρνονται οι αποφάσεις ε, και στα Ηνωμένα Έθνη πλην του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ΦΑΟ. Γίνονται λοιπόν εκτενείς διάλογοι μέχρι να καταλήξουμε σε συνένεση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, το 1994 η ΦΑΟ εξέδωσε κάποιες οδηγίες που αφορούν το δικαίωμα στην διατροφή, ώστε ο καθένας να έχει δικαίωμα στις ε, διατροφή. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο πρέπει ο καθένας να μπορέσει να το θεσπίσει στη χώρα του και να το μεταφέρει στην αρχή την νομοθεσία. Όλοι υπέγραψαν τότε, αλλά μόνο σήμερα καμιά πενταριά χώρε το έχουν εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί λοιπόν ο ΦΑΟ, αν θέλετε, να δώσει μια όθηση, αλλά τίποτε περισσότερο. Και ίσως όταν έρθει ο Γενικός Πρόεδρος, ο κ. Βρατσιάνο, θα σας πει ποια είναι η δική του αντίληψη και η άποψη για να μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποιες προτάσεις και πολιτικές. Εγώ πρέπει να σας πω επίσης ότι για εργάζομαι για να επιτεχθεί αυτή η συνένεση. Θα προσπαθήσω τώρα να δώσω κάποια στοιχεία σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε και πώς εργαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα, για να απαντήσω με στο όλο και αυξανόμενο πρόβλημα εξασφάλισης ειδών διατροφή, διατροφής για τον κόσμο, όλο δεν υπάρχει μία λύση, αλλά μία σειρά λύσεων. Πρώτα απ' όλα, την κατασπατάληση των ειδών διατροφής να την αποφύγουμε. Και είναι διπλή αυτή. Πρώτα απ' όλα, εσείς αναφέρατε κατασπατάληση εκ μέρους των πλουσίων χωρών. Είπαμε ότι 40 με 30% των ειδών διατροφή δεν πηγαίνουν στο στόμα των καταναλωτών. Υπάρχει όμω και μια άλλη κατάσταση Διαφορετική φύση. Μιλώ για την έλλειψη έργων υποδομή στι αναπτυσσόμενε χώρε. 30 με 40%, πολλέ φορέ ακόμη και ποσοστό 50% σε κάποιε χώρε τη παραγωγή στι χώρε αυτέ δεν μπορεί να διατεθεί στι αγορέ ή στο στόμα του καταναλωτή, διότι λείπουν τα έργα υποδομή τα οδικά δίκτυα, τις οργάνωση των παραγωγών, οι συνθήκες αποθήκευσης των τροφίμων κτλ. Πέραν λοιπόν από την υποστήριξη που δίδεται για να παράγουν οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, προϊόντα και να βοηθούνται οι παραγωγοί τους, είναι απαραίτητο να μπορέσουν να γίνουν και νέα έργα υποδομής. Στην περιοχή του Κέρτης θα πρέπει στα πλαίσια ε, επίσης της ισότητας ανδρών γυναικών να εξασφαλίσουμε την ισότητα και έχουμε συνειδητοποιήσει ότι 40% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Αφρική ε, είναι γεωργικές ε, ε, εκμεταλλεύσεις στις οποίες δουλεύουν γυναίκες και οι δικές τους οι γεωργικέ εκμεταλλευσει έχουν παραγωγικότητα 30% χαμηλότερη από ό,τι αυτές που, ε, στις οποίες δουλεύουν ε, οι άνδρες. Για ποιο λόγο δουλεύουν λιγότερο, όχι, αλλά έχουν πιο δύσκολη πρόσβαση στα κανάλια τα οποία θα εξασφαλίσουν ε, καλύτερα λοιπάσματα, καλύτερα μηχανήματα κτλ. Εάν λοιπόν ήταν τα πράγματα διαφορετικά, περισσότερο από 150 εκατομμύρια Αφρικανοί θα είχαν περισσότερα είδη διατροφής. Δεύτερο, το λάθος, πολιτικό ή όχι, το οποίο γίνεται στα πλαίσια τη ανάπτυξη και 30-40 χρόνια, όπου ελέγχεται ιδιαίτερω στην Αφρική. Παράγεται βιομηχανικά ηδη ή βασικά αγαθά. Για να έχετε πρόσβαση στις ε, παγκόσμιες αγορές, αν παράγετε φτωχά, κάποια στιγμή απέβει λανθασμένο. Διότι όταν αλλάζει η πολιτική των τιμών, όταν αλλάζει η τιμή των βιομηχανικών προϊόντων, δεν υπάρχει πρόσβαση στις χώρες. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει τώρα η ΦΑΟ είναι να μπορέσει να δώσει σε όλους οι οποίοι βρίσκονται επί τόπου την δυνατότητα και την ικανότητα να παράγουν. Διότι πρέπει να σας πω ότι από το ένα δις άτομα παγκοσμίως που ε, είναι σε κατάσταση ένδυας, οι 700 είναι γεωργοί. Ένα άλλο θέμα που αναφέρθηκε, η διαθεσιμότητα των γεών και η χρήση των γεών. Βεβαίως, η προτεραιότητα για τη ΦΑΟ, και το καταλαβαίνουμε, είναι να κάνει ώστε οι καλλιεργήσιμες γεές να είναι οι κατάλληλες για τη γεωργία. Γιατί? Διότι χρειαζόμαστε όλων των ειδών τη γεωργία. Εάν επιτύχουμε την ανάπτυξη σε κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες, δεν σημαίνει ότι το εμπόριο ε, ειδών διατροφής θα σταματήσει, δεδομένου ότι υπάρχουν χώρες που εξαιτία της ε, γης τους και των κλιματικών συνδικών τους δεν μπορούν να παράγουν κάποια προϊόντα, αλλά το εμπόριο ειδών διατροφής θα είναι πάντα απαραίτητο. Τώρα, ο ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός σε θέματα εγγύου ιδιοκτησίας. Πού βρισκόμαστε. Είμαστε στη μέση μεταξύ των συζητήσεων των γενικών γραμμών για τη χρησιμοποίηση της εγγύου ιδιοκτησίας και σε ένα μήνα θα επανέλθει η Επιτροπή μόνιμη για τέτοιου θέματα ε, σε συζήτηση αυτών των θεμάτων και εκεί στην Επιτροπή αυτή προσωπούνται 180 κράτη και μετά από τις προτάσεις που θα κάνει και τις αποφάσεις που θα λάβει θα πρέπει οι αποφάσεις αυτές να μπορέσουν στα πλαίσια αυτών των γενικών γραμμών να μεταφερθούν σε κάθε εθνική νομοθεσία. Τρίτον. Δεύτερον, χρήση των γεών για τη γεωργία ή για μη γεωργικές χρήσεις. Μιλούμε για βιοενέργεια. Σήμερα όντως είναι δύσκολο να ζητήσει κανείς σε χώρες που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα αυτό τη στιγμή που το πετρέλαιο έχει φτάσει τα 100 δολάρια. Όταν εγώ ήμουνα πρόεδρος της FNSA e στην Γαλλία, η τιμή του πετρελαίου ήταν 30 40 δολάρια και μου έλεγαν δεν θα είναι αποδοτική αυτό. Τη στιγμή όμως που έχει φτάσει η τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πολύ θετικό. Τώρα, πάντα από την Γεωργία είχαμε ε, την ε, παραγωγή κάποιας ενέργειας για τη βιομηχανία. Ο κύριος Γκρατσιάνο είπε τα βιοκαύσιμα έχει καλώς, αλλά χωρίς επιδότηση. Διότι αν συγχρόνως επιδοτούμε την ε, γέες μας για την καλλιέργεια βιοκαυσίμων και δεν μπορούμε να παράγουμε σε αυτές τις σε ανταγωνιστικά προϊόντα έχουμε πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να βρεθούν οι μηχανισμοί για να μπορέσει να περιοριστεί η ανάπτυξη αυτού του είδους της γεωργίας για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Τρίτο σημείο. Πώς μπορούμε να ελέγξουμε το κατά πόσο οι διάφορες γεωργικές παραγωγές μπορούν να διατηρηθούν και να διατηρηθούν. Μου θέθηκε η ερώτηση όσον αφορά τον το θέμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Έχουμε κάνει πάρα πολλές κοινέ μάχες από ό,τι φαίνεται στο εξωτερικό. Γιατί, διότι η Γεωργία και στα πλαίσια της διατροφής, ότι εγώ δεν τα διχωρίζω αυτά τα θέματα, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το κινητό τηλέφωνο και τα αυτοκίνητα Άρα είναι δύο νόμια προϊόντα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Εάν δεν έχει, χρησιμοποιείτε το κινητό σας για τρεις εβδομάδες, έχει καλός. Κάνετε καλό στην υγεία σας. Τρεις μέρες όμως ε, χωρίς φαγητό δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό. Δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει. Θίζεται και θέμα ασφάλειας. Το θέμα είναι ότι στα πλαίσια του ΠΟΕ έγινε προσπάθεια να ομοιοποιηθούν όλα τα γεωργικά προϊόντα. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Και αν θυμάστε, τελευταία φορά που πλογκαρίστηκαν τα πράγματα ήταν όταν οι Ινδιάνοι είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τους αγρότες μας, διότι θέλουμε να υπάρχει ισορροπία στους τόπους που παράγουν οι γεωργοί και ισορροπία Πιστεύω λοιπόν ότι ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δεν είναι το κατάλληλο βήμα στο οποίο μπορεί κανεί να έχει ήρεμε συζητήσει για θέματα ειδών διατροφή και ασφάλεια. Και δεν είναι τυχαίο το ότι καταλήξαμε σε αυτή την κατάσταση. Διότι εδώ και 20-30 χρόνια, στα πλαίσια του πλήρους απελευθέρωσης των αγορών, <coughs> παραγνωρίσαμε τη σημασία που έχει η παραγωγή των ειδών διατροφή και η ασφάλεια. Δυστυχώς, ε, από το 2008 και μετά, μετά από την τελευταία επιστημιστική κρίση και των προβλημάτων που δημιούργησε, πολλοί πανικοβλήθηκαν, γιατί πολλοί από τους κυβερνώντες κατάλαβαν ότι η έλλειψη τροφίμων δεν ήταν μόνο φυσικό και βιολογικό πρόβλημα, αλλά και πρόβλημα ασφαλείας για ολόκληρο τον κόσμο. Και όλοι ξέρουμε ότι ένας πεινασμένος άνθρωπος είναι επικίνδυνος επικίνδυνος που την έννοια ότι δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει, αλλά πολλές επαναστάσεις ανά τον κόσμο, εάν θέλετε, ξεκίνησαν διότι υπήρχε έλλειψη ειδών διατροφή. Σας υπενθυμίζω την Γαλλική Επανάσταση 1789 για να μην μιλήσω για την επικαιρότητα. Πολύ συχνά λοιπόν ξεχνούμε ότι η διατροφή είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των άνθρωπων. Χαίρομαι διότι στα πλαίσια του G20 και μιλώ για το G20 και όχι για το G8 διότι στα πλαίσια του G8 είχαμε πλούσιες χώρες που βοηθούσαν τις φτωχές ενώ στο G20 έχουμε πλούσιες χώρες και αναδυόμενες χώρες 20 χώρες που παράγουν το 80% των ειδών διατροφής στον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ευθύνη για όλους αυτούς και για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ και για τα αναδυόμενες οικονομίες που πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν έχουμε σήμερα την ίδια κατάσταση για να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες με αυτή που είχαμε στο παρελθόν. Παλιά ο Βορράς βοηθούσε τον Νότο, οι αναπτυγμένοι τους υποανάπτυκτους, λοιπόν, ε, ενώ σήμερα είμαστε σε κατάσταση νότου-νότου αν θέλετε έχουν αναλυθεί δεσμεύσει για να γίνει γνωστή καλύτερα η κατάσταση που αφορά την, ε, τα αποθέματα διατροφή το θέμα το επιστημιστικό ανά τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που το κάνει η ΦΑΟ για να μπορέσει να θεσπιστεί και ένα μηχανισμός πρόληψης, ώστε να μην ε, έχουμε στην αγορά ε, καταστροφικές καταστάσεις όπως αυτή που είχαμε με την πολύ μεγάλη ξηρασία στην Ρωσία και τις ε, ε, πυρκαγιές εκ των υστέρων και χρειάστηκε να κλείσουν για 15 μέρες αγορές τους οι Ρώσοι. Καταλαβαίνετε τι δημιουργήθηκε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ελέγξουμε τέτοιου είδου καταστάσεις και να τις προλάβουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις αλλαγές. Και υπάρχει ακόμη και ένα θέμα ακόμη εκρεμές, το οποίο δεν έχει επιληθεί ακόμα, είναι το θέμα των διακοιμάσεων των τιμών. Διότι και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές χρειάζονται μία κάποια ασφάλεια για να μπορέσει να, μπορέσουν κυρίως οι παραγωγοί να κάνουν τις γεωργικές του να επιβιώσουν. Κάθε φορά που υπάρχει κρίση δεν μπορούν να επιβιώσουν όλες οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Και αν κλείσει μια γεωργική εκμετάλλευση σε μια δύσκολη στιγμή, έξι μήνε μετά βελτιωθούν τα πράγματα, δεν ξανανοίγει. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τα μέσα που θα μα επιτρέψουν αυτά τα ακραία σκαμπανεβάσματα των τιμών να τα αποτρέψουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι για την διατροφή θα πρέπει να θεσπίσουμε μέτρα που να μας βοηθήσουν να περιχαρακώσουμε και να μειώσουμε την κερδοσκοπία, κυρίως την κερδοσκοπία που δεν έχει σχέση με την παραγωγή αυτή. Οι ίδιοι Αμερικανοί ήδη έχουν αρχίσει να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να μην μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Μετά από τα σκαμπανεβάσματα των ε, τιμών που είχαμε τα τελευταία χρόνια, Είδαμε ότι κοσαπλασιάστηκε η ε, η αύξηση της παραγωγής και της πώλησης δημητριακών με τόσο υψηλές τιμές. Τώρα, η κυρία Γκίνες με ρώτησε πώς μπορεί να συνεισφέρει η Ευρώπη στην διευθέτηση του προβλήματος αυτού. Σας το λέγω με σαφήνεια. Σταματήστε να κατακαιρματίζετε και να καταστρέφετε την ΚΑΠ. Είναι εξαιρετική η εμπειρία που κάναμε εδώ και 50 χρόνια με την ΚΑΠ, διότι γίναμε αυτάρκες, έχουμε μηχανισμούς ε, και δίκτυα ασφαλείας και για τα αποθέματα και για τους γεωργούς και έχουμε σταθερότητα των τιμών για τον καταναλωτή. Πρέπει να το πούμε και αυτό που ήταν ένας από τους πρώτους δικαιούχους της ΚΑΠ και από αυτούς που υποφελήθηκαν από την ΚΑΠ. Αυτό δεν είναι ε, το ίδιο για όλους, αλλά η ΚΑΠ μας βοήθησε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα θετικά στοιχεία τα οποία μας προσέφερε αυτή η πολιτική και συνδυασμένη με την περιφερειακή ανάπτυξη μπορεί να μας βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Δεύτερον, θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ΚΑΠ να συμμετέχουμε στην παγκόσμια ισορροπία όσον αφορά την ε, διατροφή. Η Ευρώπη ποτέ δεν θα μπορέσει να θρέψει αν θέλει τώρα τον κόσμο, αλλά είναι εγγυητής, διότι είναι η περιοχή του κόσμου που είναι πιο σταθερή και προσφέρει τις περισσότερες εγγύσεις. Δεν έχουμε καταστροφές, είμαστε ε, σε κατάσταση ειρήνης, μπορούμε να θρέψουμε όλους τους δικός μας τους Ευρωπαίους καταναλωτές παρά το γεγονός ότι και εμείς εισάγουμε μεγάλες ποσότητες. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε αυτοί που είμαστε. Πρώτον λοιπόν, πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Εγώ πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά από τον Ιούνιο ήμουν ένας από αυτούς οι οποίοι ήταν κατά ε, των προβλημάτων που έχουν οι δικοί μας οι φτωχοί στην Ευρώπη. Καλό είναι να λέμε θέλουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες και φτωχές χώρες, αλλά πρέπει τους φτωχούς, τους δικούς μας ανθρώπους ε, να επιβιώσουν, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και πρέπει να κάνουμε και τα δύο πράγματα συγχρόνως. Γιατί έτσι βλέπω εγώ την Ευρώπη. Τρίτη παρατήρηση. Όπως είπα και προηγουμένως, η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο συνεκτική. Δηλαδή, σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να λέει μέσα σαφήνεια ποιες είναι οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές της οι πολιτικές. Αυτά τα οποία λέγομαι για την ε, διασπάθηση και την κατασπατάληση των ε, ειδών διατροφής δεν πρέπει να τα λέμε μεταξύ μας, θα πρέπει να τα λέμε και παρά έξω. Δεν σας αποκρύπτω ότι το 42% του προϋπολογισμού μας που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση είναι κάτι που δεν ακούγεται πολύ. Πρώτα ακούμε της ΕΠΑ, τον Καναδά, τις άλλες ασυντικές χώρες και μετά... Εγώ δεν λέω ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα, αλλά πολιτικά θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Και κάτι άλλο, συγγνώμη που σας το λέω εδώ πέρα, θα μου πείτε ε, ότι δεν έχασε το παλιό του συνδικαλιστικό τεμπεραμέντο, διότι εγώ συνδικαλιστής ήμουνα στο παρελθόν για πολλά χρόνια. Άκουσα να λέτε προηγουμένως για το ρόλο των αγροτών στην, ε, ε, για το περιβάλλον, ε, γιατί ξέρετε ότι οι χωρικοί καμιά φορά βλάπτουν το περιβάλλον αλλά μετά το επανορθώνουν και λέτε ότι θα πρέπει όλα αυτά να μπουν στο, στην καρδιά της προβληματικής ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν εμείς όμως δεν κρατήσουμε τους χωρικούς την επικράτειά τους, αν τους, δεν τους πούμε «Κοιτάστε, σας έχουμε ανάγκη, μείνετε εκεί που είστε, ε, αν δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε δεν πειράζει, χωριάτες είστε εκεί καθίστε». Όχι, Όλα αυτά έχουν μία τιμή. Η τροφιμική ασφάλεια έχει μία τιμή. Και εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε και το εισόδημα των γεωργών. Όταν πάμε εμείς στην Αφρική σε ένα χωριό και τους λέμε στους νέους, κοιτάξτε, που σπουδάσανε κάτι και τους λέμε μείνετε στο χωριό γιατί σας χρειαζόμαστε. Και όταν αυτοί βλέπουν τι γίνεται ε, παρά έξω και ότι στο χωριό τους δεν μπορούν να ζήσουν, τι κάνουν, ε, εντείνουν την αστιφιλία. Το θέμα ε, τι του νερού μας ανησυχεί επίσης, επίσης το θέμα είναι να συμβάλλουμε στην προσαρμογή όλων των πληθυσμών στις αλλαγές είναι ένα θέμα με το οποίο, για το οποίο συνεργαζόμαστε και με άλλες οργανώσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ καλέστε και τον Γενικό Διευθυντή διότι αυτός θα είναι πολύ πιο στο ψαχνό της υπόθεσης. Εγώ βρίσκομαι αρμόδιος για θέματα governance για θέματα διαχείρισης και όχι για καθημερινά ζητήματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, πρόεδρε Γκριό, να στείλετε την πρόσκληση ε, της Επιτροπής μας τον Κρατσιάνο Ντεσίλβα να έρθει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συνεισφέρει και αυτό στη συζήτηση για την τροφιμική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Ε, δύο μέρες δουλέψαμε γερά. Η επόμενη συνεδρίαση είναι 6 Φεβρουαρίου στις 15 εδώ στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ, καλή δουλειά.